του Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύνθεση της δικής μας Επιτροπής έφυγε ο κύριος Καμάλ και αντικαταστάθηκε από τον κύριο Χάναν. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Καμάλ που ήταν τέταρτος αντιπρόεδρος έφυγε και γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε τώρα στην εκλογή ενός νέου αντιπροέδρου η προηγούμενη συνάντηση λοιπόν αφορούσε την εκλογική διαδικασία και για να ακούσουμε επίσης, α όχι έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα, ο ίνιγκο διαδικαστικό. Συμφωνώ να κάνουμε αυτό το οποίο λέτε για τον κύριο Κάμαλ, ο οποίος ε, δεν ήταν και πάρα πολύ παρόν, αλλά εν πάση περιπτώσει φεύγει από την Επιτροπή μας, φεύγει από την Αντιπροεδρία και εσείς τι μας προτείνετε, να προχωρήσουμε στην εκλογή κάποιου άλλου στη θέση του. Αυτό προτείνετε. Α, προτείνετε τον κύριο Χάναν απευθείας, ο οποίος δεν είναι εδώ βέβαια. Ε, θα ήθελα ο κύριος Χάνα να έρθει εδώ και να τον ψηφίσουμε, να ξέρουμε τουλάχιστον ποιο ψηφίζουμε. Είναι θέμα ευγένειας απέναντι στην Επιτροπή γιατί ε, νομίζω ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε κάποιον που να εκπροσωπεί την Επιτροπή μας αν δεν τον ξέρουμε. Εγώ δεν θα υπερψηφίσω ε, κάποιον ο οποίος δεν είναι παρόν. Δεν ξέρω, ο κύριος Ντάφο ο οποίος έχει συμμαχία με τους Βρετανούς συντηρητικού. Εγώ δεν είπα ότι θα πρέπει να εκλέξουμε. Εγώ περιορίστηκα να πω ότι η μερίσια διάταξη εγώ δεν έκανα και καμία πρόταση. Περιορίστηκα στο να πω ότι έχει αλλάξει η μερίσια διάταξη γιατί θα πρέπει επίσης να τεθεί το θέμα της εκλογής του τετάρτου αντιπροέδρου. Θα το κάνουμε αυτό εφόσον είναι εφικτό. θυμίζω ότι ε, μόνο το θέμα της εκλογικής διαδικασίας ήταν για συζήτηση αλλά μετατέθηκε το πολύ σημαντικό θέμα της τροποποίησης του άρθρου 136 της Συνθήκης και γι' αυτό είναι απαραίτητο επίσης να τεθεί και το θέμα της εκλογής του τετάρτου αντιπροέδρου. Εφόσον συμφωνείτε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη όπως διατυπώθηκε ε, μπορούμε να συνεχίσουμε. Βρισκόμαστε στο σημείο 2 στις ανακοινώσεις του Προέδρου και θυμίζω ότι στη συνάντηση των συντονιστών της 1ης ε, Φεβρουαρίου τέθηκε το θέμα των εισηγητών και η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος επέλεξε να ορίσει τον εισηγητή για τη δημοσιονομική διαδικασία για το 12. Στα πλαίσια λοιπόν της μελλοντικής διοργανικής συμφωνίας ε, και συνεργασίας στα θέματα του προϋπολογισμού. Ε, ήμουν εγώ υπεύθυνο, αλλά θα το αναλάβει άλλος αντιπρόεδρος, δεν είναι μαζί μας σε αυτή τη φάση. Νομίζω λοιπόν και ότι πρέπει να σας θυμίσω αυτά τα οποία έχουν ήδη υποθεί μετά από τη συνάντηση και κλεισμένων των θυρών τη σχετική με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κάποιοι από εμά που ήμασταν παρόντες, δεν χρειάζεται να πω πολλά, να πληροφορήσω πάντως ότι οι διαδικασίες για την ένταξη θα ολοκληρωθούν μετά από δύο περαιτέρω συναντήσεις, μία τον Μάρτιο και μία τον Μάιο. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να δημιουργήσει ένα άτυπο όργανο που να αποτελείται από εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όρισε ε, τμήμα της ομάδας αυτής τον κύριο Γκουερέρο που παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις και ε, ε, τον υποφαινόμενο. Οι πολιτικές ομάδες έχουν επίσης την δυνατότητα η κάθε μία να ορίσει ένα εκπρόσωπο. Για να πάνε λοιπόν τα πράγματα γρήγορα και όπως είπα και όπως είπε ο συνάδελφος Γκουερέρο στο προηγούμενο κομμάτι της συνάντησης Πρέπει να τα συνδυάσουμε τα πράγματα έτσι ώστε η ομάδα αυτή να αρχίσει να δουλεύει γρήγορα. Όπως είπα η διαπραγματευτική ομάδα θα συναντηθεί το Μάρτιο και το Μάιο και γι' αυτό η ομάδα αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει πριν το Μάρτιο. Λοιπόν μετά από αυτά περνάω στο σημείο 3. Το σημείο 3 είναι αυτό που δεχθήκαμε να βάλουμε στην ημερήσια διάταξη ορίζουμε λοιπόν τον τέταρτο αντιπρόεδρο μετά από την αντικατάσταση ε, του Καμάλ από τον Χανάν. Η ομάδα του Καμάλ και τον Χανάν μας είπε ότι θα προτείνει τον συνάδελφο κύριο Φόξ ο οποίος είναι παρόν εδώ εφόσον υπάρχουν και άλλες προτάσεις για τον ορισμό του κυρίου Φόξ στη διάθεσή μας. Αγαπητέ Ίνιγκο, Πολύ ευχαρίστω και ευχαριστούμε τον συνάδελφο Φόξ για τη διάθεση που έδειξε. Και είναι πάρα πολύ οικοδομητική η παρουσία του εδώ στην Επιτροπή και χαιρόμαστε να αναλάβει την Αντιπροεδρία. Εάν δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις, νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε εκλεγμένο ως τέταρτο αντιπρόεδρο, διαβοής βέβαια, τον κύριο Φόξ. Συγχαρητήρια κύριε Φόξ. Πάμε τώρα. Στο πιο σημαντικό σημείο είναι η τροποποίηση του άρθρου 136. Είναι εδώ οι συγγητές. Δίνω το λόγο στον συνάδελφο Βερχόφστατ. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που ζητώ ευθύς αμέσως το λόγο. Αλλά εγώ σε λίγο έχω μία διάσκεψη προέδρων με τον κυρίο Τρισέ για το ίδιο θέμα. Αυτό βέβαια δεν οφείλεται στη δική μας επιτροπή αλλά στη διάσκεψη των, των προέδρων. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν η μερίσια διάταξη να οργανώνεται κάπως πιο ευέλικτα ούτως ώστε κάποιος να συμμετέχει σε δύο συνεδριάσεις. Έχουμε εμείς λοιπόν συνεδρίαση για την αλλαγή των συνθηκών, μετά έχουμε διάσκεψη των Προέδρων σε 10 λεπτά για την ε, διάσκεψη των Προέδρων και διμερή των δύο εισηγητών με τον κύριο Τρισέ πάλι για την τροποποίηση των συνθηκών. Δηλαδή πρέπει να είμαστε τρισδιάστατοι. Αλλά τέλος πάντων, Είναι αδύνατο να συμμετέχει κανείς με το σωστό τρόπο στις συνεδριάσεις και ζήτησα το λόγο για να πω τη γνώμη μου. διότι στην προηγούμενη μας συνεδρίαση το συζητήσαμε ήδη το θέμα και θα το συζητήσουμε και στις επόμενες εβδομάδες εγώ μίλησα και με τον κύριο Γκουαλτιέρη και με τον κύριο Μπροκ πιστεύω όμως ότι θα είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας. Αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε θα ήθελα Ε, θα ήθελα να αρχίσω με ένα ανακοινοθέν ε, τύπου του Reuters πριν από καμιά ώρα ε, τυπώθηκε. Είναι μια ανακοίνωση του κυρίου Βέμπερ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που λένε ότι θα είναι και ο διάδοχος του κυρίου Τρισέ αλλά αυτά είναι σχετικά πράγματα γιατί όλα μπορούν να συμβούν στο μεταξύ διότι μόνο όταν σας διορίζουν πραγματικά από εμπειρία δηλαδή ε, είστε όντως διορισμένος όλοι τα ξέρουμε αυτά έτσι έχουν τα πράγματα στην πολιτική τι λέει τώρα αυτό το ανακοινοθέν που έσκασε μύτη πάνω κάτω πριν από δύο ώρες να το διαβάσω στα αγγλικά γιατί από το Reuters έρχεται οπότε φυσικά είναι στα αγγλικά οι προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις ε, στα μέσα του προπολογισμού της Ένωσης δεν είναι αρκετά φιλόδοξες και αφήνουν πάρα πολλά στις κυβερνήσεις. Είπε ο Άξελ Βέμπερ τη Δευτέρα στέλεχος ε, της Κεντρικής Τράπεζας και συνεχίζει μια γαλλογερμανική συμφωνία επέφερε κάποιες αλλαγέ καθώς το Παρίσι επέμενε να υπάρχει περισσότερη πολιτική υποπτία από τις χώρες ε, κάτι το οποίο θα μπορούσε να καθυστερήσει η διαδικασία ε, λήψη αποφάσεων παρόμοια με το σημερινό σύστημα και συνεχίζει λέγοντας και λέει ότι γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε το πακέτο ε, που έχουμε στο τραπέζι. Αυτό όμω δεν είναι δική μα δουλειά, είναι δουλειά τη ΕΚΟΝ από ό,τι φαίνεται. Αλλά γιατί όμως είναι και δική μας δουλειά. Διότι ο κύριος Βέμπερ λέει και ο Chief Economy, ο κύριος Στάρκ και ο κύριος Τρισέ λένε όσοι δηλαδή είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του ευρώ λένε ότι το πακέτο που κατέθεσε η Κομισιόν στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν δεν αρκεί. Το ξέρουμε αυτό γιατί οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πριν από δύο μέρες άρχισαν να εργάζονται για τη συνέχεια. Άρχισαν να εργάζονται επί ενός δευτέρου πακέτου οικονομικής διαχείρισης. Δηλαδή πρέπει να δημιουργηθεί και Οικονομική Ένωση και ε, παράλληλα δίπλα στην Νομισματική Ένωση που δεν έχει νόημα να είναι μόνη της. Εμείς λοιπόν ε, ως Κοινοβούλιο έχουμε επίσημα, έξι προτάσεις, τέσσερις είναι με συναπόφαση. Και θα πρέπει να εκφραστούμε λοιπόν για αυτές και πρέπει να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Αλλά τι λέει ο κύριος Βέμπερ, όπως είπε και ο κύριος Στάρ και ο κύριος Τρίσε, ότι το πρόβλημα με το πακέτο είναι ότι το Συμβούλιο, δηλαδή τα κρατη πρέπει να δώσουν το ok πριν μία διαδικασία για υπερβολικό έλλειμμα ξεκινήσει από την Κομισιόν συμπεριλαμβανομένων και των κυρώσεων. Αυτό είναι και το δύνατο σημείο του πακέτου. Γιατί, Γιατί το Σύμβουλιο βασιζόμενο στα άρθρα 121 και 126 της συνθήκης λέει ότι πρώτα πρέπει το Συμβούλιο να αποφασίσει για υπερβολική ελληματική θέση πριν αποφασίσει η Κομισιόν για τις κυρώσεις και πριν βρεθεί και η ειδική πλειοψηφία η οποία μπορεί να μπλοκάρει αυτές τις κυρώσεις που θα έχει αναλάβει η Κομισιόν. Όλοι λοιπόν θεωρούν ότι αυτή είναι η αδυναμία του πακέτου που έχουμε στο τραπέζι. Διότι στο παρελθόν εγώ 9 χρόνια τα όλα αυτά Μια-δυο φορές είχα τη δυνατότητα να αντιμετωπίσω αυτά τα προβλήματα και είδαμε ότι υπήρχαν χώρες οι οποίες δεν σεβόντουσαν το σύμφωνο σταθερότητα, αλλά δεν ξεκινούσε καμιά διαδικασία εναντίον τους γιατί το Συμβούλιο δεν αποφάσιζε για να τους, ε, βάλει μέσα στη, να τους εντάξει στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος όπως ε, απαιτούσαν οι συνθήκες. Εντάξει, αφήστε που πρέπει να αλλάξει και το σύμφωνο σταθερότητα και όλα αυτά, αλλά αυτά θα είναι στη συνέχεια. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Το Κοινοβούλιο και η Οικονομική Νομισματική λένε ότι αρχίζουν να το σκέφτονται και λένε αυτά πρέπει να λειτουργούν αυτόματα, δεν χρειάζονται ή αυτοματισμοί. Ή αυτόματες θα είναι οι κυρώσεις ή δεν θα είναι αυτόματες. Αλλά αυτά τα αυτόματα μέτρα δεν, δεν μπορούν να υπάρχουν. Όπως όταν κάποιος είναι έγκυος ή είσαι έγκυος ή δεν είσαι έγκυος. Εγώ προσωπικά δεν έχω εμπειρία εγκυμοσύνης, αλλά αυτό τέλος πάντων ξέρετε δεν μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, η ιδέα ποια είναι. Πρέπει να ενισχύσουμε το πακέτο και αυτό ε, κυριαρχεί στην οικονομική νομισματική τώρα. Και έχουμε δύο δυνατότητες. Ή μπορεί αυτό να είναι εφικτό μέσα στα πλαίσια της τωρινής συνθήκης βάσει του άρθρου 133. Το άρθρο 133 της συνθήκης λέει σαφώς ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο από κοινού και χωρίς ε, παρεκκλήσεις των αρμοδιοτήτων της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορούν με την ε, τακτή διαδικασία να αναλάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη χρήση του ευρώ. Ένας καλός δικηγόρος θα συνηγορούσε υπέρ αυτού. Θα έλεγε λοιπόν να έχουμε το άρθρο 133 και βάσει του άρθρου 133 αυτοματοποιούμε το πακέτο της οικονομικής διαχείρισης και κάνουμε και ένα βήμα προς τα μπρος. Δεν είμαστε εμείς που θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, η εικόνα θα την κάνει, αλλά μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας στους συναδέλφους μας. Δεύτερη δυνατότητα, και γι' αυτό το συζητάω εδώ, Έχουμε άλλοι που, είναι άλλοι που λένε ότι το 133 δεν φτάνει γιατί το 133 αφορά μόνο σε τεχνικά μέτρα. Για να δώσουμε λοιπόν πραγματικό αυτοματισμό στις κυρώσεις χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό από το 121 και 126. Χρειάζεται μια προσθήκη λοιπόν. Σε ποιο άρθρο? Μα, στο 136 πάλι, γιατί το 136 είναι αυτό που μιλάει για την Ευρωζώνη. Και αυτό θέλω να ρωτήσω, να ζητήσω από τον κύριο ε, Μπρόκ και τον κύριο Γκουαλτιέρη να βάλουν μέσα στην έκθεσή του. αυτό το σημείο. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί μέσω της ΕΚΟΝ ότι πρέπει να ενισχύσουμε και να κοινωνικοποιήσουμε τις κυρώσεις της οικονομικής διακυβέρνησης ή θα, πρέπει να κάνει μια ευρύ ερμηνεία του άρθρου 136 ή θα πρέπει να θέσει μία προσθήκη στο άρθρο 136 το οποίο εμείς ε, συζητάμε στην Επιτροπή μας διότι πρέπει να γνωμοδοτήσουμε για το θέμα. Αυτό είναι το συγκεκριμένο μου ερώτημα ε, γιατί θεωρώ ότι εδώ πρέπει να γίνει στην Επιτροπή μας στη φάση δηλαδή που οι δύο οι εισηγητές μας ε, συντάσσουν την έκθεση. Βασίζομαι λοιπόν στους κυρίους Τρίσε, Σταρκ και Βέμπερ, όλους αυτούς του διαχειριστές του, του ευρώ που λένε ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν τώρα, για τον ίδιο το μηχανισμό. Ο μόνιμος μηχανισμός που θέλουμε να δημιουργήσουμε με την τροποποίηση του άρθρου 136. Ζητώ στην έκθεση Μπροκ Γουαλτιέρη να υπάρξει μία διατύπωση που να επιτρέπει και είτε την διακυβερνητική εφαρμογή του μηχανισμού είτε την κοινοτική εφαρμογή του μηχανισμού. Εμείς θα μπορούσαμε να βρούμε μία διατύπωση, μια φρασεολογία που θα αφήνει ανοιχτό το θέμα. Εάν το γράψουμε όπως λέει το Συμβούλιο, τότε εμείς θα παραμείνουμε στην διακυβερνητική χρήση του μηχανισμού. Αλλά εμείς ως μέλη της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων θα πρέπει να προτείνουμε μια διατύπωση που θα δίνει τη δυνατότητα να ερμηνεύουμε το μηχανισμό διπλά και διακυβερνητικά και κοινοτικά διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η κοινοτική μέθοδος είναι η καλύτερη μέθοδος για να διαχειριστούμε αντίστοιχους μηχανισμούς. Ζητούμε λοιπόν να γίνει χρήση των λέξεων κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπεται και η κοινοτική ε, μέθοδος στο μηχανισμό σταθερότητας. Δεύτερη παρατήρηση κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Γκουαλτιέρη και ο κύριος Μπρόκ στην έκθεση τους αναφέρουν ένα άλλο πρόβλημα που ακόμη δεν έχει ρυθμιστεί και το πρόβλημα που δεν έχει ρυθμιστεί να το πούμε βέβαια είναι αυτή η μάχη που χάσαμε για τον προϋπολογισμό του 2011 πρέπει να ξανασυζητήσουμε για τον ρόλο που θα πρέπει να παίζει το Κοινοβούλιο στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί να μην αναφέρουμε λοιπόν και αυτή την ιδέα που κυκλοφόρησε και που θεωρώ ότι είναι μια ιδέα, καλή ιδέα του κυρίου Λαμασούρ που παρουσίασε ως πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών και ζήτησε να γίνει μια διάσκεψη ε, <coughs> το 2012, μια διάσκεψη μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου, Κομισιών και Εθνικών Κοινοβουλίων για τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ένωσης. Αυτή θα ήταν μια επιθυμία που θα μπορούσαμε να εκφράσουμε στην έκθεση. Αυτές ήταν οι τρεις παρατηρήσεις μου και ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά κύριε Πρόεδρε που θα είμαι τόσο αγενής και θα φύγω αλλά γιατί, θα φύγω γιατί έχουμε την διάσκεψη των Προέδρων η οποία συνεδριάζει για το ίδιο θέμα με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαριστώ κύριε Βερχόφστατη για αυτήν την τόσο πυκνή τοποθέτηση. Κρίμα που δεν είναι εδώ οι συγητές Γουαλκέρι και Μπρόκ, αλλά ε, βρίσκονται σε άλλες επιτροπές. Μας είπαν ότι θα είναι εδώ στις 4, τέλος πάντων. Εμείς καταγράφουμε την τόσο σημαντική σας τοποθέτηση και καταγράφουμε επίσης ότι δεν θα μπορεί δεν θα μπορείτε να βρίσκεστε ταυτόχρονα σε δύο επιτροπές διότι η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων απαγορεύει την κλωνοποίηση ως εκ τούτου δεν μπορείτε να έχετε αυτήν τη διπλή διάσταση. Ο κύριος Μέντες Δεβίγο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση είναι σημαντική. Διότι οι συγητές αυτής της Επιτροπής, της Θεσμικής Επιτροπής, είναι οι συγητές της Επιτροπής. Δεν εκφράζουν δηλαδή μόνο τον εαυτό τους, πρέπει να εκφράζουν το κοινό αίσθημα της Επιτροπής μας. Οπότε όταν θα έρθει η ώρα της σύνταξης αυτής της έκθεσης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις γνώμες των πολιτικών ομάδων. Οι μαζί μας ζήτησαν σε όλους τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων να τους στείλουμε ένα κείμενο που να εκφράζουμε το τι θέλουμε να περιέχει αυτή η έκθεση. Οι σοσιαλιστές το κάνανε, το κάνανε οι ΕΛΚ και μάλιστα προς μία γραμμή που συγκλίνει προς τις θέσεις του κυρίου Φερχόφστατ. Πιστεύω λοιπόν ότι θα προσφέραμε σε αυτές τις στιγμές μέσα σύγχυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσφέραμε λοιπόν χρηστές υπηρεσίες σε αυτή τη φάση δηλαδή που τα γεγονότα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα και όπου είχε η Κομισιόν υποβάλει προτάσεις κατάλληλες για το Σεπτέμβριο, και όταν τις εξετάζουμε το Φεβράριο είναι πια ξεπερασμένες από τα γεγονότα. Πρέπει λοιπόν εμείς να ξεπεράσουμε αυτές τις, ε, να υπερβούμε αυτές τις προτάσεις. Αυτά δηλαδή προς, προς τα εκεί τίνουν αυτά που μας λέει ο κύριος Βερχόφστα, ο κύριος Βέμπερ, ο κύριος Τρισέκ, ακόμη και με το Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας. Δείτε αυτό το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σαρκοζή. Προβλέπουν πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν την, την οικονομική διακυβέρνηση αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο των έξι μέτρων που πρότεινε η Κομισιόν. Πιστεύω λοιπόν εγώ για την έκθεση Μπρόκο Γουαλτιέρη ότι θα πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτο, να απαντήσουμε σε αυτό που μας ρωτάνε. Δηλαδή, να εκτιμήσουμε ναι ή όχι αν συμφωνούμε με την τροποποίηση του άρθρου 136 της συνθήκης. Και αυτό με μια τροποποίηση που συνοδεύεται και από μια πρόταση τροποποίησης. θα δούμε τι προτάσεις ε, θα προκύψουν, ε, θα μας τις υποβάλει και η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά. Ταυτόχρονα όμως εμείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκθεση ως μέσο για να ορίσουμε το πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης που θέλουμε. Πρέπει λοιπόν εμείς να ξεπεράσουμε τα γεγονότα. Λέτε εσείς ότι, λέμε μάλλον ότι τα γεγονότα ξεπέρασαν τις προτάσεις της Κομισιόν. Ε, και εμείς λοιπόν να ξεπεράσουμε τα γεγονότα. Παράδειγμα. Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με την αξιολόγηση των προσχεδίων προϋπολογισμών των κρατών μελών με τους μεγάλους προσανατολισμούς για οικονομικά ζητήματα και λέω εγώ και για κοινωνικά έτσι όπως έχουν τοποθετηθεί σήμερα Ενηχεύουν κινδύνους διότι όπως τα λέγαμε και στα ισπανικά και στα ελληνικά διατρέχουμε τον κίνδυνο να μετατραπούν όλα αυτά σε ένα ένα μπλα μπλα μπλα Πρέπει λοιπόν εμείς να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκθεση για να πούμε ακούστε. Όταν εδώ έχουμε μία πρόταση της Κομισιόν για ένα προσχέδιο προϋπολογισμού οποιοδήποτε κράτος μέλους που πάει προς τη λάθος κατεύθυνση, δεν θα πρέπει εμείς να, να, να αντιδράσουμε με ένα ψήφισμα γενικό, πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση και το κράτος που δεν θα ακολουθήσει, ε, δεν θα κάνει τίποτα, θα πρέπει να υποστεί συνέπειε. Δεν μπορούμε εμείς να εξετάζουμε, να, να υποπτεύουμε το εξάμεινο και μετά στο τέλος να λέμε «Α, η τάδε χώρα δεν ακολούθησε τις συστάσεις μας». Αυτό εγώ εννοώ ως ξεπέρασμα της υπάρχουσας κατάστασης. Και μετά έχουμε και τη συζήτηση που έχουμε κάθε μέρα στις εφημερίδες για τα ευρωομόλογα, τα ευρωσεκιούριτις όλα αυτά θα πρέπει να τα βάλουμε μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο. Τι είδους ευρωσεκιούριτις έχει, τι τύπου θα είναι. Δεν θα μπορούσαμε εμείς μέσω αυτών των ευρωομολόγων να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα και τα σχέδια και οτιδήποτε άλλο, όχι μόνο μπόνους για την είναι ε, επιχορηγήσει του κρέους. Όλα αυτά λοιπόν τα πακέτα, Euro Securities, έξι νομοθετικά πακέτα της 22ης Σεπτεμβρίου που μας τα δώσει η Κομισιόν. Αυτά αποτελούν ένα καλό πλαίσιο για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε τις πίστες που θέλουμε να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Και αυτό μέσω της έκθεσης Brock και Γκουαλτιέρη. Αφού άκουσα και τον κύριο Γκουερέρο και τον κύριο Νταφ, πιστεύω ότι και αυτοί τείνουν προ την ίδια κατεύθυνση αυτών που λέω κι εγώ. Και ξανάρχομαι στην αρχή της τοποθέτησή μου. Εμένα μου φαίνεται ότι θα ήταν καλό ο κύριος Μπροκ και Γκουαλτιέρη να εντάξουν στο κόρπους της έκθεσής τους όλες αυτές τις προτάσεις. Εγώ νομίζω ότι αυτή θα ήταν μία διανοητική και πολιτική συνεισφορά πολύ σημαντική. Διότι αυτό το συζήτησαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Συμβούλιο και το Μάιο πάλι θα το ξανασυζητήσουμε. Και δεν μπορούσαμε εμεί να είμαστε πάντα ουραγοί αυτών που να αποφασίζουν τα άλλα, τα, τα ευρωπαϊκά όργανα. Πιστεύω λοιπόν, πρόεδρε, ότι πρέπει να καταστεί σαφέ ότι η ομάδα μου θέλει στην έκθεση Μπροκ Γκαλγουελτιέρη να έχουμε όχι μόνο την ερώτηση συμφωνείτε με το 136 τροποποίησή του και κατά αυτόν τον τρόπο τον άλλον, αλλά να συμπεριλαμβάνονται και οι γενικέ γραμμέ τη οικονομική διακυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Μέντε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μόλις τώρα ήρθε ο κύριος Γκουαλτιέρη, περιμένουμε και τον κύριο Μπροκ. Θα ήθελα να καθησυχάσω τον συνάδελφο Γκουαλτιέρη που ήταν απόν και δεν άκουσε τις παρεμβάσεις ε, υψηλού περιεχομένου των κυρίων κυρίων Ντεβίγκο και Φερχόστατ. Η γραμματεία μας όμως κράτησε τα πρακτικά και θα του μεταφέρει και γραπτά αυτά τα οποία ακούστηκαν. που να πάρετε μια ανάσα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Γκουερέρο και μετά θα δούμε ακριβώς την σειρά των ομιλητών και θα σας δώσουμε το λόγο. Ο κύριος Γκουερέρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ περιεκτική η τοποθέτηση του κυρίου Φερχόστατ. Αλλά ο κύριος Φερχόστατ μας είπε ότι ήδη ήρθε σε επαφή με τον κύριο Γκουαλτιέρη και με τον κύριο Μπρόκ και ότι στα πλαίσια αυτής της συνεδρίασης ε, που έχουν σήμερα με, τους ε, με τη διάσκεψη των Προέδρων και με τον κύριο Τρισέ οι εισηγητές θα έχουν ε, τη δυνατότητα να ακούσουν χοντρικά αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Βερχόφστατ. Άκουσα τα αυτά που μας είπε ο κύριος Μέντες Δεβίγο. Τρεις πολιτικές ομάδες, ο κύριος Μέντες Δεβίγο, εγώ και ο κύριος Νταφ, στείλαμε στους εισηγητές ε, μερικές σκέψεις ε, γενικού χαρακτήρα για την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης. Σκέψεις που όπως είπε και ο κύριος Μέντες Δεβίγκο καλό θα ήταν να συνοδεύουν την έκθεση. Γουαλτιέρη και Μπρόκ. και να μην περιορίζεται να λέει συμφωνούμε ή διαφωνούμε με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όμως θέλω να επισημάνω ότι διατρέχουμε έναν κίνδυνο. Δηλαδή, να φανταστούμε ότι όλες οι τροποποίησεις οι απαραίτητες για την οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να ερμηνεύονται και συνταγματικά. Να το πω αλλιώς όπως υπόθηκε και στην προηγούμενη συζήτηση. Όχι απλώς εμείς έχουμε ένα πακέτο προτάσεων για την οικονομική διακυβέρνηση, αλλά όσο περνάει ο χρόνος προβάλλει ένα συνεχές κατεπήγον που απαιτεί προτάσεις, νέες προτάσεις. Μας το έδειξε αυτό και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση αναβρασμού. Ε, υποβάλλονται προτάσεις, ε, μέτρα, διότι συμπεραίνουμε ότι τα τρέχοντα μέτρα ή αυτά που ελήφθησαν στο παρελθόν δεν επαρκούν για να εγγυθούν την οικονομική διακυβέρνηση μέσα στην Ένωση και τη σταθερότητα του ευρώ. Πρέπει όμως να είμαστε και επαρκώς ακριβείς για να κάνουμε διάκριση μεταξύ ρύθμισης της οικονομικής διακυβέρνησης και συνταγματικής ερμηνείας της οικονομικής διακυβέρνησης. Με ποια έννοια το λέω. Μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική συνένεση στην οικονομική, επί της οικονομικής διακυβέρνησης και, όχι τόσοι επί των συνταγματικών τροποποίησεων. Και είναι επικίνδυνο να ξεκινήσουμε εμείς ε, βρείτε, τα μεταρρυθμίσεις της, ε, του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και να μην είναι τόσο ευρέως αποδεκτές. Όπως είναι και η θέση των εισηγητών να τοποθετηθεί η Επιτροπή μας επί του ερωτήματος που μας τίθεται για την τροποποίηση του άρθρου της συνθήκης. Γιατί η η θέση του κυρίου Φερχόφστατ με οδηγεί να σκεφτώ ότι θα μπορούσε να ανοίξει τους ασκούς του αιώλου για την τροποποίηση της συνθήκης και αυτό με επιβαρυντικές πολιτικές επιπτώσεις. Ε, ευχαριστώ. Οργανώσαμε αυτή τη συζήτηση αφήνοντας να τοποθετηθούν οι συνάδελφοι πριν από τους εισηγητές. Οι εισηγητές βέβαια μπορούν να τοποθετηθούν μετά. Ρωτώ, κανένας άλλος βουλευτής θέλει το λόγο, ο Χέφνερ. Ναι, περίμενα, γιατί θεώρησα λογικό, εφόσον δεν είχαμε γραπτό σχέδιο έκθεσης, να μιλήσουν οι συγητές. Να μας πούν που βρίσκονται. Τα είπαν αυτά την τελευταία εβδομάδα, αλλά υπέρχαν κάποιες διαφορές σε αυτά τα οποία μας είπαν οι δύο εισηγητέ. Πριν επαναλάβουμε λοιπόν αυτά τα οποία συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ ήθελα να ακούσω του εισηγητέ και μετά να τοποθετηθώ. Οι συγητές γύρω από το θέμα αυτό έχουν, ε, ε, οφείλουν να είναι παρόντες και σε άλλη συνάντηση και δυστυχώς γι' αυτό δεν είναι μαζί μας. Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, και εγώ κάτι παρόμοιο. Θεωρώ πως η συζήτηση έδειξε πως αυτό το οποίο συζητήσαμε την τελευταία φορά φαίνεται ακόμη πιο αντιφατικό σήμερα. Γι' καλό θα ήταν να μας πούν τώρα ό,τι έχουν να μας πούν οι συγητές, γιατί ακούγοντας αυτά τα οποία ακούσαμε και λαμβάνοντας πόσο και την επιστολή του κυρίου Μόν από την Ευρωπαϊκή ε, Ομοσπονδία Συνδικάτων να δούμε πώς θα έχουμε σε αυτή την κατάσταση την ευρύτερη δυνατή συζήτηση και στα ζητήματα ουσίας και στα ζητήματα τύπου για την αλλαγή της συνθήκης και μετά θα ήθελα να τονίσω πως η θέση μας την οποία παρουσίασαμε την προηγούμενη φορά νομίζω πως είναι η κατάλληλη διέξοδος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους εισηγητές. Ποιος θα, προ... θα μιλήσει πρώτος, ο Γκουαλτιέρη πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη και εξ ονόματος του Μπροκ. Ήμασταν προσκεκλημένοι στην Επιτροπή Προϋπολογισμών σε μια συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό, η οποία αντίθετα από ό,τι είχε προβλεφθεί καθυστέρησε και δεν ήμασταν σε θέση να φύγουμε βέβαια πριν κλείσει ο πρόεδρος Λαμασούρ γιατί στράφηκε και σε μας και δεν μπορέσαμε να φύγουμε έγκαιρα. Άκουσα ένα τμήμα των παρεμβάσεων, μου δόθηκαν κάποια στοιχεία, όχι λεπτομερή, κάποιον από τις ιδέες που δεν μπορέσαμε να ακούσουμε. Να πω ότι αυτά τα οποία συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα αποδεικνύουν πόσο δίκιο είχαμε όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση αυτή και όταν υποχραμίζαμε ότι πίσω από αυτό το θέμα, το σχετικά τεχνικό θα έλεγα, το της προσαρμογής της συνθήκης δηλαδή, με μια νέα πρακτική η οποία βρίσκεται εξελίξη, κρύβεται περισσότερο κάτι άλλο κρύβεται μια εξέλιξη θα έλεγα ταραχώδης των πολιτικών και οικονομικών και θεσμικών διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία όπως συχνά γίνεται σε περιπτώσεις επιτάχυνσης της ιστορίας τα θετικά και τα αρνητικά της εξέλιξης ε, αναμειγνύονται και συγχέονται και οι συνδυασμοί ανάμεσα στις δύο αυτές πλευρές επηρεάζουν τις ισορροπίες τις οποίες θα καταλήξουμε. Εγώ θεωρώ προσωπικά θετικό το ότι υπήρξε μια όθηση προς μια στενότερη οικονομική συνεργασία και διακυβέρνηση. Ταυτόχρονα ανησυχώ όταν διαβάζω στα έγγραφα τα οποία ποτέ δεν κατετέθησαν βέβαια επίσημα και τα οποία βρισκόντουσαν ε, σαν βάση της συζήτησης στο μηχανισμό ενός μηχανισμού παραλλήλου με τους αντίστοιχους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται ένα νέο Eurostat και προβλέπεται επίσης και ένα, ένα νέο φόρουμ κοινοβουλευτικό των χωρών που συμμετέχουν σε αυτήν τη νέα συνεργασία εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, νέες αντιτιθέμενες μεταξύ τους πρωτοβουλίες Επαναλαμβάνω ότι εγώ δεν επανέρχομαι στα θέματα στα οποία είχα την δυνατότητα να εκφράσω την προηγούμενη φορά, θέματα που έχουν σχέση με το ρεαλισμό που θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει και που τον γνωρίζουν οι συνάδελφοι που με γνωρίζουν. Να τονίσω μόνο κάποιες συνταγματικού χαρακτήρα αντιρρήσεις γύρω από το ότι η πρότασή μου η οποία παρουσιάζει μια κάποια διαφοροποίηση της νέας φράσης η οποία προστίθενται στην Παύλα 1 σε σχέση με την Παύλα 3 της συνθήκης και η οποία αυξάνει για ορισμένους τις αρμοδιότητες της Ένωσης. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είμαι πεπισμένος ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει αύξηση των κοινοτικών αρμοδιοτήτων, και είναι κάτι το οποίο είναι θα έλεγα συμβατό με την διαδικασία της απλοποιημένης αναθεώρησης. Και εδώ θα συμφωνήσω και με τον κύριο Γκουερέρο ότι η ιδέα του να ξεκινήσει τώρα ένα νέο εργοτάξιο διοργανικό γύρω από τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι κάτι το ε, ιδιαίτερα μη ρεαλιστικό. Πάντως πρέπει να ληφθούν κάποιες τέτοιες αποφάσεις οι οποίες ε, μπορεί να ληφθούν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικά με το λεγόμενο σύμφωνο της ανταγωνιστικότητας ε, θα ήθελα να παρασέμψω στο 136 της Συνθήκης της Λισαβόνας το οποίο επιτρέπει να κάνουμε ακριβώς αυτά τα οποία προβλέπονται με τις ίδιες εγγυήσει, αλλά όλα αυτά στο εσωτερικό της διοργανικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αυτό να οδηγεί ή να απαιτεί μια εξωτερική της Ένωσης συμφωνία. Συμφωνώ βέβαια ότι μια, ένα τέτοιο σύμφωνο θα μπορούσε να ενταχθεί ή να μην ενταχθεί στο χώρο του 133. Αυτό είναι μια επιλογή που είναι υποσυζήτηση. Από τον τρόπο λοιπόν με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε εμείς το θέμα της μεταρρύθμισης της συνθήκης μπορεί να επηρεάσουμε ελπίζω <coughs> αυτές τις διαφορετικές και διαφοροποιούμενες αντιφάσεις μερικές φορές οι οποίες χαρακτηρίζουν τα, τα κοινοτικά πράγματα τον τελευταίο καιρό. Ελπίζω λοιπόν ότι μέσω μιας νέας ρύθμισης και καθορισμού των στόχων είτε θα είναι πιο φιλόδοξη είτε θα είναι πιο ρεαλιστική Παρ' όλα αυτά θα πρέπει εμείς να συνδυάσουμε λόγω του ευαίσθητου ε, του, ε, του προβλήματος να εντείνουμε το κοινοτικό χαρακτηριστικό, να αντιμετωπίσουμε τον διακυβερνητικό κίνδυνο και να μην, ε, και να μην κενώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από το ίδιο της το μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Μπρόκ. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ακόμα. Από το τέλος της περαμένης εβδομάδας πλέον έχουμε να κάνουμε με τρία ζητήματα. Πρώτα απ' όλα είχαμε την αλλαγή της συνθήκης και την ομοθεσία, το Σύμφωνο Σταθερότητας. Τώρα, με τη δέσμευση του Συμβουλίου της Παρασκευής, μιλάμε και για ένα σύμφωνο ανταγωνιστικότητας. Όλα αυτά σχετίζονται σε έναν βαθμό από τη σκοπιά της Επιτροπή μας αυτό που είναι το λιγότερο προβληματικό είναι το ζήτημα του Συμφώνου Σταθερότητας. Καθώς ε, βεβαίως ρυθμίζονται ξεκάθαρα τα τη συμμετοχής των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και έχει δικαίωμα συναπόφασης το Κοινοβούλιο. Εντάξει, το πώς θα γίνει λοιπόν είναι με τη φυσιολογική πολιτική διαδικασία. Μετά έχουμε δύο τομείς δηλαδή το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας και την αλλαγή της συνθήκης και δεν ξέρουμε πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα θεσμικά. Γιατί μέχρι τώρα νομίζαμε πως είναι κάτι το διακυβερνητικό και συζητήσαμε την τελευταία φορά για την πίεση που υπάρχει ε, για να μην έχουμε δυσκολίες αγορές 27 Μαρτίου όταν θα έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να είμαστε διατεθειμένοι για συμβιβασμούς. Δεν ε, ξέρω τώρα τι γίνεται με το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας. Από τη μία έχουμε τα έγγραφα που προέρχονται ε, από την χώρα μου, όπου θέλω να αναφέρω το εξής. Όταν οι εκπρόσωποι ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων προσκαλούνται, θα έχουν στόχο τον συντονισμό της ανταγωνιστικότητας και εκτός ε, της εθνικής ε, νομοθεσίας. Για Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίποτα, κανένα λόγος. Και εδώ πέρα πρέπει να ομολογήσω πως εδώ έχουν αρχίσει να χτυπάνε τα καμπανάκια. Να χτυπάς να γερμός. Θέλω να επαναλάβω πως η αλλαγή της συνθήκης είναι αναγκαία γιατί και για νομικούς και για πολιτικούς στόχους για να οδηγηθούμε γιατί ξέρετε πως θα μπορούσαμε να πάμε σε... στο να αποτύχει αυτός ο μηχανισμός σταθερότητας δηλαδή ενώπιον του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου και μετά να έχουμε πάει σε μια καταστροφή. Και βέβαια είμαστε και περιορισμένοι από πλευρά χρόνου, αλλιώς θα πάμε σε καταστροφή 27 Μαρτίου. Αλλά από την άλλη κοιτάω τέτοια έγγραφα τα οποία ζητάνε από τη μία ευθύνη και από την άλλη μιλάνε μόνο για κράτη-μέλη. Οπότε πρέπει να έχουμε κάποιες διευκρινήσεις ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ποια είναι τα ωφέλη της αλλαγής της συνθήκης αλλά και την εμπλοκή όσον αφορά την κυβερνητική ε, διαδικασία για το σύμφωνο ανταγωνιστικότητα. αν και εγώ θεωρώ πως στο άρθρο 136 παράγραφος 1 υπάρχουν όλα τα, αρμο, τα σχετικά για ένα σύμφωνο ανταγωνιστικότητα. Μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της ε, συνθήκης. Γνωρίζω πως κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι επίσης ε, στη χώρα μου, του οποίου γνωρίζω, έχουν επίσης την ίδια άποψη. Γι' αυτό θα ήθελα να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις στην έκθεσή μας. Κάνουμε μία έκθεση στην οποία ε, περιέχεται ένα ναι, τίποτα παραπάνω. Και μάλιστα ένα πακέτο το οποίο αντιμετωπίζει τα ζητήματα συνολικά. Αλλά εγώ θα ήθελα να έχουμε μία πρόταση που θα ξεχαρίσει αυτά τα ζητήματα που σας είπα πριν να αποφασίσουμε στην Ολομέλεια. Και αν δεν έχουμε διευκρινίσει από το Συμβούλιο, ε, καλά, τότε δεν ξέρω και εγώ τι θα συμβεί. Αλλά επειδή ξέρουμε όλοι την προθεσμία της 27 η Μαρτίου, ίσως να έχουμε κάποιες ε, διευκρινήσει. Νομίζω έτσι έχουν τα πράγματα. Εγώ και ο κύριος Γκαλτιέρη συζητήσαμε και με τον κύριο Τρισέ, με τον Παρόσο την προηγούμενη εβδομάδα και τον Φαν Ρόμποϊ. Ο Φαν Ρόμποϊ είπε παρακαλούμε να τα συζητήσετε αυτά τα ζητήματα αλλά βεβαίως ε, οι άλλοι μας είπαν και ποια είναι τα πολιτικά τους όρια λένε πως οι πολιτικές μας επιθυμίες ε, Ε, δηλαδή το να πάμε στην παράγραφο 136 τα λοιπά δεν ε, ισχύουν. Επίσης άλλε χώρε ανέφεραν που στέλνουν δημοψήφισμα γιατί έχουμε μετάβαση αρμοδιοτήτων. Λοιπόν, χρειαζόμαστε απλοποιημένη διαδικασία, πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν τα δημοψηφίσματα, έχουμε την 27 Μαρτίου ω μια επικίνδυνη ημερομηνία και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τις συζητήσεις και ακούγοντας βέβαια και τις δηλώσεις του πρόεδρου της Κομισιόν του κυρίου Μπαρόσο στην ε, Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω πως ξαφνικά και αυτός ανησυχεί για το τι θα γίνει με τα θεσμικά όργανα της ε, κοινότητας. Βεβαίως αυτός ανησυχεί περισσότερο για την Κομισιόν και όχι για το Κοινοβούλιο, αλλά νομίζω πως έχουμε έναν καλό ε, συνομιλητή όταν μιλάμε για τα διακυβερνητικά ζητήματα και το κατά πόσον θα επικρατήσει αυτή η αντίληψη. Οπότε όπως σας είπα δεν έχουμε καταλήξει ακόμα οριστικά, ούτε εγώ, ούτε ο κύριος Γκαλτιέρη θα συναντηθούμε και με τον κύριο Τρισέξανα να δούμε τι ιδέες θα προκύψουν για να καταλήξουμε σε μια πρόταση που θα σας κάνουμε αλλά εγώ βλέπω πως θα κινηθούμε προς μια τέτοια κατεύθυνση ε, δηλαδή να μην αποκλείουμε τίποτα γιατί όπως σας είπα έχουμε και αυτό τον Ιωνί έτσι, συνταγματικό χαρακτήρα των θεμάτων αυτών. Ε, Κανένας δεν σήκωσε το χέρι του για να στήσει το λόγο. Α, Χέμπνεχ. Ναι, ευχαριστώ τους δύο εισηγητές για την διατύπωση της, της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε όλοι. Δεν ξέρουμε ακόμα πού θα καταλήξει αυτή η πορεία. Με μεγάλη ανησυχία λοιπόν παρατηρώ σε αυτή τη σύντομη συζήτηση δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε πως έχουμε μια οπισθοδρόμηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και εδώ πέρα βεβαίω αναφέρομαι στη δημοκρατική εξέλιξη της Ευρώπης γιατί θεωρώ πως ειδικά με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο ευρώ είναι αναγκαίο να εξελίξουμε την κοινοτική μέθοδο και όχι να πάμε ακόμη πιο πίσω. Αυτό θα πρέπει να είναι ο κοινό μας στόχος και σε σχέση με το Συμβούλιο θεωρώ πως ε, αποστολή της έκθεσής μας και του Κοινοβουλίου και πρωτίστως της Επιτροπής μας είναι να εκφράσουμε την άποψη του Κοινοβουλίου ως ε, του μέρους εκείνου που εκφράζονται οι πολίτες της Ευρώπης. Δηλαδή να ενισχύσουμε την κοινοτική μέθοδο, να έχουμε στο δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υποστηρίζω λοιπόν αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γκουαλτιέρη, την πρόταση περί μετατροπής αυτής της παραγράφου 3 στο προτινόμενο κείμενο και ενσωμάτωσής της στην παράγραφο 1. για να δημιουργηθεί έτσι, να δοθεί ένα μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Τώρα δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί δεν έχουμε και κάποια πρόταση μπροστά μας. Νομίζω πως και οι δύο εισηγητές πρέπει να ζητήσουν εξ ονόματος της Επιτροπής μας να μην, να μην πράγματα όπως έχει, γιατί εδώ πέρα πρέπει να γράφονται εξελίξεις για το πώς και στο μέλλον θα αντιμετωπίσουμε στο πολιτικό επίπεδο τέτοια ζητήματα και πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ευχαριστώ. Μπορούμε λοιπόν να ολοκληρώνουμε με αυτό το σημείο γιατί έχουμε ακόμη ένα σημαντικό σημείο. Περνάει και ο χρόνος. Ευχαριστώ τους εισηγητές. οι οποίοι συγκλίνουν με τις θέσεις της Επιτροπής μας και θα τα πούμε στις 17 του μηνός στην ε, έκτακτη συνεδρίαση και ελπίζουμε ότι θα λυθεί αυτό το τόσο πολύπλοκο μαθηματικό ζήτημα. Α, 14 του μηνός και όχι 17. Έκανα λάθος, έκανα λάθος. 14 του μηνός ε, θα συναντηθούμε σε έκτακτη συνεδρίαση με αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη στο Στρασβούργο. Διορθώνω λοιπόν 14 Φεβρουαρίου θα ξανασυζητήσουμε το θέμα. Πάμε τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Πρόταση αλλαγής του κανονισμού για την ε, εκλογή με απευθείας με καθολική ψηφοφορία των Ευρωβουλευτών. Έγινε μια διάσκεψη σχετικά στο Κέμπριτζ. Είναι παρόν εδώ ο καθηγητής Γκρίμετ. ο οποίος και εκπροσωπεί δηλαδή και όλους τους υπόλοιπους μαθηματικούς που συμμετείχαν στο σεμινάριο του Κέμπριτζ. Δεν ξέρω αν ο κύριο Νταφ θέλει να κάνει εισαγωγή, να δώσουμε κατευθείαν το λόγο στον καθηγητή Γκρίμετ. Νομίζω πω καλό είναι να μιλήσει πρώτα ο κύριο καθηγητή και μετά να λάβω εγώ το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, έχετε τον λόγο κύριε καθηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με προσκαλέσατε. Είναι χαρά μου να είμαι εδώ ως μαθηματικός. Πρώτα απ' όλα να πω στα μέλη της Επιτροπής σας βεβαίως πως ε, είμαι πιο συνηθισμένος να μιλάω στους φοιτητέ μου παρά σε ευρωβουλευτές και ξέρω πως θα με προσγειώσετε στην πραγματικότητα εάν πάω στη λάθος κατεύθυνση. Το περασμένο Σαββατοκυριακό μια ομάδα μαθηματικών μετά από πρόσκληση της Επιτροπής σας συναντήθηκε στο Κέμπριτζ και συζήτησε επί δύο ημέρες την κατανομή των εδρών μεταξύ των κρατών μελών. Τα προσωρινά μας ευρήματα νομίζω τα έχετε ήδη και νομίζω θα δείτε στο γραφείο σας κάποιες σελίδες που προβάλλονται και στην οθόνη. Είναι δύσκολο ίσως να δει κανείς στην οθόνη. Λοιπόν, λέγομαι Τζέφρι Γκρίμετ, ε, καθηγητής ε, στατιστικής ε, στο Κέμπριτζ οι μαθηματικοί, όπως ξέρετε, προσπαθούμε να είμαστε λογικοί, αφαιρετικοί, να ξεκινήσουμε από κάποιες αρχές. Αυτές λοιπόν οι προσωρινές μας συστάσεις, ε, αυτά τα οποία βλέπετε σήμερα δεν θα αλλάξει, αλλά η τελική μας ακόμα έκθεση δεν ε, έχει ολοκληρωθεί. Υπήρχαν αρκετοί μαθηματικοί οι οποίοι επιλέγησαν για την εμπειρογνωμοσύνη τους στον τομέα αυτό από πολλές χώρες και πανεπιστήμια και μας ε, συμβούλευσε ένα μέλος του Πανεπιστήμιου του Αμπαντίν για ζητήματα πολιτικής και βεβαίως ήταν παρόντες όχι μόνο μέλη της επόμενης γενιάς αλλά και πρόσωποι της Επιτροπής σας ε, τους οποίους ευχαριστούμε που ήρθαν. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ε, κάναμε αυτά τα οποία μας ζητήσατε και τίποτα παραπάνω, οπότε η έκθεσή μας και τα συμπεράσματά μας περιορίζονται στην εντολή μας. Εάν θέλει η Επιτροπή να μας δώσει βεβαίως διαφορετική εντολή, ευχαρίστως να το εξετάσουμε. Αλλά η έκθεση που σας παρουσιάζω σήμερα σχετίζεται με την εντολή την οποία λάβαμε από την Επιτροπή σας μέσω του εισηγητού. Σας υπενθυμίζω το σημείωμα που μοίρασε πριν από λίγες εβδομάδες ο κύριος εισηγητής όταν είπε πως ε, στόχος συνάντησης ήταν να συζητήσουμε και να προτείνουμε ή δυνατόν ένα μαθηματικό τύπο. Εγώ τα έχω υπογραμμίσει αυτά που βλέπετε εκεί πέρα τονίζω το μαθηματικό τύπο, για την ανακατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάποιες λέξεις κλειδιά. Ο τύπος πρέπει να είναι διαφανής. Φαντάζομαι διαφανής όχι μόνο σε πολιτικούς ή μαθηματικούς, αλλά σε, στον κόσμο. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να διατηρηθεί αυτός ο μαθηματικός τύπος και σε πιθανές αλλαγές στα θεσμικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Και υπάρχει παράγραφος που αφορά τον στόχο να σταματήσει το πολιτικό παζάρι και να είναι στιβαρές κάποιες αλλαγές που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά όσον αφορά τη μετανάστευση και τις δημογραφικές αλλαγές και βεβαίως τη διεύρυνση μέσω των νέων κρατών μελών. Οπότε οι περιορισμοί οι συγκεκριμένοι που έχουμε εδώ πέρα σε αυτή την έκθεση είναι οι εξή. Πρώτα απ' όλα, το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 751 βουλευτές. Μας είπαν πως δεν ανάγκη να είναι 751 ή και 750 ή μπορεί να είναι και 520 ακόμα, αλλά βεβαίως θα προξενούσε έκπληξη σε κάποιους αν ε, δεν ήταν ε, τουλάχιστον αν δεν πλησίαζε ή ήταν ίσο με το 751 ο αριθμός. Κατόπιν, είχαμε ένα ελάχιστο όριο 6 εδρών. Κανένα κράτο μέλο δεν θα είχε λιγότερο από 6 ευρωβουλευτέ. Τρίτον, κανένα κράτο μέλο δεν θα πρέπει να έχει πάνω από 96 έντρε. Έχουμε ανώτατο και κατώτατο όριο. Και. Μετά βεβαίω κάποια εσωτερική συνέχεια, δηλαδή να μην έχει κάποιο μικρότερο κράτος περισσότερες έντρες από μεγαλύτερη χώρα, φυσικό. Και τέλος η κατανομή να κάνει σεβαστή τη λεγόμενη φθήνουσα αναλογικότητα. Οπότε έγινε κάποια συζήτηση για τη φθήνουσα αναλογικότητα και το πώς θα ερμηνευτεί. Και σας αναφέρω από την εκθέση του 2007 των κυρίων Λαμασούρ και Σεβερίν στις σημειώσεις τους αναφέρω συζητούν την αρχιτεκτονική δομή της Ένωσης, συζητούν κάποιες αρχές και λένε πώς θα προχωρήσουμε εντός αυτού του πλαισίου. Η ιδεώδης εναλλακτική λύση βεβαίως θα είναι να συμφωνήσουμε σε ένα μαθηματικό τύπο φθήνουσας αναλογικότητας που βεβαίως θα άντεχε και σε μελλοντικέ αλλαγές λόγω διεύρυνση δημογραφικών αλλαγών. Όπως βλέπετε εδώ πέρα μαθηματικός τύπος που δεν θα αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας. Ίσως ζητάμε πάρα πολλά. Και μετά έκαναν μία πρόταση σύμφωνα με την οποία βεβαίως ε, κάθε, πιο, κάθε βουλευτής πιο πολυπληθούς κράτους θα εκπροσωπεί περισσότερους ανθρώπους από βουλευτές από μικρότερα κράτη. Άρα όσο πιο μεγάλο το κράτος τόσο περισσότεροι ψηφοφόροι αντιστοιχούν σε κάθε βουλευτή. Υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα με αυτή την ερμηνεία που πρέπει να συζητήσω πριν σας δείξω τα βασικά, τις βασικές μας συστάσεις. Το θέμα είναι, όταν θα συζητήσουμε τις διάφορες μεθόδους κατανομής των εδρών, ε, είναι πως υπάρχουν δύο φάσεις όσον αφορά τους μαθηματικούς τύπους. Πρώτα απ' όλα είναι να ορίσουμε αρχές και να διαρρέσουμε τον αριθμό με τον άλλον και έτσι καταλήγουμε σε μια θεωρητική κατανομή εδρών. Αλλά βεβαίως είναι... αυτό οδηγεί σε δεκαδικού αριθμού. Δεν μπορεί να είναι το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει 69,3 βουλευτέ μα το έχει πει ο εισηγητή αυτό. Οπότε αυτό το 69,3 πρέπει να στρογγυλοποιηθεί. Οπότε πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε μια στρογγυλοποίηση των αριθμών σε ακέραιους. Όπως ξέρετε η στρογγυλοποίηση γίνεται με διάφορους τρόπους το θέμα της ρογγυλοποίησης παραδείγματο χάρη έχει απασχολήσει πάρα πολύ το ζήτημα το ανάλογο στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ε, κατανέμονται οι έδρες των πολιτιών στην Γερουσία και στην ε, Βουλή των Αντιπροσώπων. Και υπάρχουν βεβαίως και οι συνέπειες της τρογγυλοποίησης. Η αναπάντεχη συνέπεια βεβαίω ε, του αυστηρού ορισμού τη έκθεση ε, Λαμασούρου Ρεβεσούν είναι πως εάν κάνουμε αυτή τη στρογγυλοποίηση μετά παραβιάζουμε την αρχή αυτή του τύπου. Και αυτό φαίνεται σε πάρα πολλέ λογικές πιθανέ ε, κατανομές. Θα δούμε κάποια παραδείγματα αργότερα. Από μαθηματική σκοπιά ε, αναζητούμε αποφάσεις βεβαίως με βάση κάποιες αρχές και μας είπαν να αποφύγουμε καταστάσεις ε, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολιτικά παζάρια ή καυγάδες. Ε, βεβαίως το πρόβλημα είναι πως υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με αυτόν τον κανόνα, είναι πως υπάρχουν θεωρητικές ευρωπαϊκές ενώσεις και θεωρητικά μεγέθη κοινοβουλίων για τα οποία δεν υπάρχει λύση που θα ικανοποιεί αυτή τη συγκεκριμένη ερμηνεία της θήνουσας αναλογικότητας. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση για αυτή την Ευρώπη ή για την επόμενη αν θέλετε. Για την παρούσα ή την επόμενη. Έχουμε μια πρόταση λοιπόν την οποία ε, ελπίζουμε να δείτε με θετικό μάτι. Μιλάμε λοιπόν για μια ελαφριά αλλαγή αυτής της ερμηνείας και ο λόγος τον οποίο υπολογίζουμε, ε, που θυμάστε ότι είναι ο πληθυσμός δια της έδρας, αντικαθίσταται από τον θεωρητικό λόγο την αναλογία πριν τη στρογγυλοποίηση. Προτείνουμε δηλαδή την ε, προσθήκη πέντε μικρών λέξεων που λέει πως ο λόγος πριν προχωρήσουμε στρογγυλοποίηση σε ακέραιους αριθμούς θα ικανοποιεί αυτή την αρχή της θύνουσας αλλαγωγικότητας. Και δεν είμαστε νομικοί, αλλά θεωρούμε πως αυτό είναι εντών, εντός ε, των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, καθώς η νομοθεσία επιτρέπει κάποιες μικρές αποκλήσεις ή τέλο πάντων κάποια διατύπωση θα το επιτρέπει αυτό. Εάν υιοθετήσετε, γιατί είπα αν ευθύσουμε τέλο πάντων μαθημένο ω καθηγητή, εάν υιοθετήσετε αυτή την πρόταση θα τα κάνει αυτά πιο εύκολα για του μαθηματικού, καθώ όλα τα συστήματα τα οποία εξετάσαμε για να δώσουμε μία απάντηση με ένα μαθηματικό τύπο ικανοποιούν την ε, πρόταση Cambridge αλλά όχι την ερμηνεία Λαμασούρη Σεβερίν για να ε, προλάβω κάποιε συζητήσει. Κανένα από του δύο ορισμού δεν είναι πιο ε, ισχυρός ισχυρό από τον άλλον. Δηλαδή, έχουμε κατανομέ που ικανοποιούν την πρώτη και όχι τη δεύτερη προπόθεση, οπότε δεν ξέρω αν κάποιο είναι πιο ισχυρό από τον άλλον. Τώρα, γιατί το, το κόκκινο εδώ πέρα στις διαφάνειες αυτές σημαίνει κίνδυνο. Ποιος είναι λοιπόν ο κίνδυνος εδώ πέρα έχουμε ένα δεδομένο μέγεθο του Κοινοβουλίου και υπάρχει βεβαίω κάποιο κίνδυνο να μην καταλήξουμε σε λύση. Και αυτό προκύπτει γιατί έχουμε καταστάσεις όπως ε, η σημερινή όπου κάποια κράτη-μέλη έχουν παρόμοιου πληθυσμού. Θα, ε, μπορώ να μιλήσω γι' αυτό αργότερα αν ενδιαφέρεται κάποιο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τα τρία επίθετα που ήταν στην εντολή μας. Δηλαδή, διαρκής, διαφανής και αμερόληπτη η λύση. Διαρκής όσον αφορά δηλαδή τις πιθανές αλλαγές στην ε, θεσμική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μακροπρόθεσμα. Διαφανής δηλαδή να μπορεί να εξηγηθεί με μια απλή και λογική εξήγηση και βεβαίως αμερόληπτη όσον αφορά την ε, πολιτική τοποθέτηση. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν πως ε, ήμασταν μαθηματικοί και ε, ήμασταν οπωσδήποτε αμερόληπτοι όσον αφορά την καταγωγή και την πολιτική τοποθέτηση. Βεβαίως αυτοί οι περιορισμοί δεν μπορούν να ορίσουν το σύστημα. Και όπως παρατηρήσατε στο παρελθόν υπάρχουν πολλές λύσεις ε, σε αυτό το πρόβλημα που πληρώνουν αυτές, αυτούς τους περιορισμούς. Για να πάμε λοιπόν παραπέρα πρέπει να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις για την τρέχουσα κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς θα εξελιχθεί για να δούμε το τι σημαίνει βιωσιμότητα. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27 κράτη-μέλη, το μικρότερο έχει πληθυσμό 400.000, το μεγαλύτερο έχει ένα πληθυσμό 200 φορές περισσότερο. Μιλάμε για μια, ένα τεράστιο φάσμα. Οι μελλοντικέ ε, τώρα εντάξει δεν θα πω εγώ ποιες θα είναι, χωρών, αλλά οπωσδήποτε θα συμπεριλάβουν μικρές χώρες και μακροπρόθεσμα θα είναι και μεγαλύτερες χώρες. Θα υπάρχει μετανάστευση και δημογραφική αλλαγή. Αυτό συμβαίνει και σήμερα, συνέβη και στο παρελθόν, συνέβη πέρυσι και θα συνεχίσει να συμβαίνει. Οπότε οποιαδήποτε νούμερα και κατανομή σας δείξω παρακάτω, σέβονται βεβαίως πλήρως τα νούμερα της Eurostat, αλλά ε, όχι βεβαίως το πραγματικά νούμερα επτόπου. Τέλος, εμείς έχουμε ένα κουτάκι αν θέλετε, στο οποίο μπαίνουν οι αριθμοί και από το οποίο βγαίνει η κατανομή. Τα νούμερα λοιπόν αυτά είναι αυτά τα οποία βρήκαμε στο site της Eurostat. Οπότε η πρότασή μας είναι να υιοθετήσουμε ένα σύστημα το οποίο εμείς λέμε βάση συν αναλογικότητα. Βασιστήκαμε λοιπόν στα επίθετα που ορίζουν τους περιορισμούς και εξετάζοντας την τωρινή και πιθανή μελλοντική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε πως έχουμε ένα στιβαρό και διαφανές ε, σύστημα για την κατανομή ε, μελών, μεταξύ μεδρών μεταξύ των κρατών μελών βάση πρώτα απ' όλα. Έχουμε ένα σταθερό αριθμό που πάει στο κάθε κράτος μέλος. Αυτός ο αριθμός λέγεται βάση. Η βάση εδώ πέρα ορίζεται ως B. Ο αριθμός B βεβαίως Έχουμε 27 καρατιμέλη, 27 μπι, αν το αφαιρέσουμε από το, από το 751 αφήνει έναν αριθμό εδρών μη κατηλημένων και αυτές οι έδρες μετά κατανέμονται αναλογικά σύμφωνα με τον πληθυσμό των κρατών μελών. Βεβαίως η ζωή δεν είναι ποτέ τόσο απλή γιατί έχουμε κάποιους περιορισμούς για το μέγιστο και τον ελάχιστο αριθμό. Ο ελάχιστος είναι το μπι, η βάση και βεβαίως υπάρχει και ε, το μέγιστο μέγεθο του Κοινοβουλίου. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν αλγόριθμο για να έχουμε αυτού του περιορισμούς. Ο κλασικός τρόπος, ο οποίος είναι ελκυστικός και αυτόν, βεβαίω ε, προτείνουμε να ακολουθήσουμε, είναι βεβαίω να βρούμε έναν διαιρέτη. Ορίζουμε λοιπόν εναντί τον διαιρέτη, που θυμάστε είπαμε έχουμε το B e επί 27, και έχουμε τις υπόλοιπες θέσεις και μετά ο διαιρέτης σημαίνει ένα μέγεθος ψηφοφόρων ή πληθυσμού που αντιστοιχεί αναβουλευτή. Ο διαιρέτης λοιπόν έχουμε και μετά τον πληθυσμό, οπότε ο οποίος, αντικα... Ε, ο οποίος αντικατοπτρίζεται από το οπότε π διαντί είναι ο αριθμός ανδρών. Π διαντί λοιπόν είναι ένα κλάσμα και δεν μπορούμε να έχουμε βεβαίως βουλευτές δεκαδικούς, πρέπει να στρογγυλοποιηθεί. Οπότε πρέπει να συζητήσουμε πώς θα γίνει η στρογγυλοποίηση. Οπότε όπως σας είπα έχουμε πίδι αντί εντός αγγυλών. Και θα καταλήξουμε σε κάποια μέθοδο για τη στρογγυλοποίηση. Οπότε έχουμε βάση συν αυτόν τον αριθμό αντί. Εάν αυτό ξεπερνά το μέγιστο αριθμό 96, τότε το αντικαθιστούμε από το μέγιστο, το 96. Έχουμε ανώ όριο. Οπότε το σύστημα αυτό κατανέμει έδρες στα διάφορα κράτη-μέλη και βεβαίως αν το πει είναι σταθερό το D ε, εξακολουθεί να κυμαίνεται και δεν ξέρουμε πόσες έδρες θα έχουμε συνολικά. Οπότε παίζουμε τώρα με το D μέχρι το συνολικό μέγεθος του Κοινοβουλίου ταυτιστεί με τον προκαθορισμένο αριθμό. 751 αυτή τη στιγμή δηλαδή, σύμφωνα με την εντολή που μας δώσατε. Αυτή είναι η γενική δομή ενός ε, συστήματος που θεωρούν πως είναι εύρωστο και διαφανές. Επίσης, και αυτό δεν είναι εντός εντολής μας, μπορούσαμε να το δούμε ως έναν τρόπο να διακρίνουμε μεταξύ κράτους και πολίτη. Τα κράτη έχουν ένα αριθμό εδρών και οι υπόλοιπε έδρε κατανέμονται σύμφωνα με τον πληθυσμό. Οπότε, αν και δεν ήταν στην εντολή μας, όπως σας είπα, λαμβάνουμε υπόψη μας την δήλωση πως ε, πρέπει αυτός να είναι ένας δίκαιος τρόπος ε, κατανομής των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θεωρούμε πως είναι εύκολο να δείξουμε με διάφανο τρόπο το ότι αυτή η μέθοδος είναι δίκαιη για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίω, υπάρχουν κάποιοι νούμεροι, κάποια αριθμοί εδώ πέρα, δηλαδή κυρίως η βάση και η μέθοδος στρογγυλοποίησης. Οπότε ε, να δώσω την απάντηση και μετά να δείτε γιατί ισχύουν αυτοί οι περιορισμοί. Εμεί προτείνουμε λοιπόν μετά από τη συζήτησή μα να οριστεί η βάση στο 5 και η στρογγυλοποίηση να είναι προ τα πάνω. Οπότε οποιοδήποτε κλάσμα, οποιοδήποτε δεκαδικό στρογγυλοποιείται προ τα πάνω. Εφόσον κάθε κράτο μέλο δεν έχει βεβαίω μηδενικό πληθυσμό, αλλιώ δεν θα χρειαζόταν και ευρωβουλευτέ, πάντα έχει ένα θετικό αριθμό εδρών και άρα τουλάχιστον παίρνει μία παραπάνω. Με τη στρογγυλοποίηση, με το συνδυασμό αυτών των δύο κανόνων έχουμε έξι τον ελάχιστο αριθμό εδρών και νομίζω τρία κράτη-μέλη, τρία μικρά κράτη-μέλη με αυτό το σύστημα έχουν έξι έδρες. Οπότε δύο πράγματα έχουμε εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα συζητήσαμε τον τύπο της προσέγγισης και όπως σας είπα μπορώ να σας πω αργότερα για το πώς καταλήξαμε σε αυτό το σύστημα αλλά αυτά θα υπάρχουν στην οριστική μας έκθεση. Αυτό το οποίο σας παρουσίασα λοιπόν είναι η βάση. Μπορείτε να μας πείτε γιατί δεν είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη. Θεμητή ερώτηση. Μετά, Υπάρχουν τρεις ε, πολύ φυσικοί τρόποι στρογγυλοποίησης, προς τα κάτω, μετά το να πάμε προς τον πλησιέστερο ακέραιο, 5,4 δηλαδή σημαίνει 5, 5,6 σημαίνει 6, αλλά το 5,5 το συζητάμε, αλλά σπάνια βρισκόμαστε στο 5,5. Και βεβαίως υπάρχει στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Να πάμε προς τον πλησιέστερο ακέραιο προς τα πάνω. Οπότε έχουμε δύο επί τρεις επιλογές. Τι κάνουμε με την εντολή μας. Μικρότερη βάση ευνοεί τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη γιατί αφήνει μετά περισσότερες έδρες να διανεμηθούν. Και κατά αναλογία με τον πληθυσμό παίρνουν περισσότερες έδρες τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη. Μεγαλύτερη βάση, αντιστρόφως, ευνοεί τα μικρότερα κράτη. Γιατί έχουν κάποιον αριθμό που λαμβάνουν το ή και μετά κατά αναλογία προς τον πληθυσμό. Η στρογγυλοποίηση λοιπόν. Ε, γενικά είναι πιο αποδεκτό πως ε, η στρογγυλοποίηση προς τα κάτω ευνοεί τα μεγαλύτερα κράτη, η στρογγυλοποίηση προς τα πάνω τα μικρότερα. Δείτε το ως εξή. Εάν ένα κράτος έχει π.χ. 60,1 έδρες ε, έχει 60. Η, ανα... η αναλογία δηλαδή ε, έχει, πολύ, έχει πολύ λίγο αλλάξει. Εάν όμως έχει 6,1 και πάρει 7, ε, είναι πολύ μεγαλύτερη. Παίρνει αναλογικά πολύ περισσότερες έδρες. Οπότε ευνοούνται με την στρογγυλοποίηση προς τα πάνω τα μικρότερα κράτη. Το να στρογγυλοποιήσουμε προς τον πλησιέστερο ακέραιο θεωρείται λίγο πολύ ουδέτερο σε σχέση με το μέγεθο του κράτους μέλους. Οπότε ο συμβιβασμός των μαθηματικών του Cambridge. Για να σας υπενθυμίσω πως είμαστε και μαθηματικοί. Υπάρχουν τρεις παράμετροι. Ο ελάχιστος αριθμός κατά κράτος, ανά ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να χωρέσει το κοινοβούλιο. Ας πάρουμε το π αγγλικό, είναι ο πληθυσμός μιας χώρας. Αν το διαιρέσουμε με τον διαιρέτη, το μετατρέπουμε σε ακέραιο και το προσθέτουμε στη βάση. Αυτή, αυτό είναι το θεωρητικό σχήμα το οποίο μπορεί να χαρακτηρίσει ένα κράτος. Αλλά μπορούμε να πάρουμε και το μη. Το μη, το εμ είναι το maximum. Αν προσθέσει κανείς το S με το σύνολο των μελών του Κοινοβουλίου, δεν φτάνει κανείς στον μέγιστο αριθμό. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε την ρύθμιση που θα μας επιτρέψει στο να καλύψουμε τον συνολικό αριθμό των μελών που επιτρέπεται στο Κοινοβούλιο. Βλέπετε το μικρό M λοιπόν, ο ελάχιστος αριθμός εδρών ανακράτος, το μη κεφαλαίο που είναι ο μέγιστος αριθμός, εδρών ανακράτος και το H λατιν, ε, αγγλικό που είναι το μέγεθος του Κοινοβουλίου. Στην τελική ε, μορφή νομίζω ότι θα δείτε και μεγαλύτερους πίνακες σχετικά με τις προτάσεις τις οποίες καταλήγουμε. Στην ουσία βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της έκθεσής μας, η οποία έκθεσή μας σχολιάζει και παρουσιάζει τους πίνακες τους οποίους σας έχουμε δώσει, 27, 28 κτλ. Καταρχάς θα πρέπει να δείτε ακριβώς πώς είναι αυτοί οι πίνακες. Βλέπετε ε, τις χώρες. Οι χώρες πηγαίνουν από μεγαλύτερη προς μικρότερη. Μετά βλέπετε ακριβώς τον αριθμό του πληθυσμού ε, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που μας έχει δώσει η Eurostat. Μετά βλέπετε το 5. Το 5 είναι ο διαιρέτης. Ξέρουμε τι είναι ο διαιρέτης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε αν εφαρμόσουμε το διαιρέτη τον αριθμό τον τελικό ο οποίος ε, δεν μπορεί να ξεπεραστεί και αφορά το σύνολο των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Αμέσως μετά έχουμε τον πληθυσμό, ο οποίος όμως έχει διαιρεθεί από τον διαιρέτη. Και εδώ έχουμε δηλαδή την θεωρητική κατανομή πέραν της βάσης. Η Ουγγαρία σαν παράδειγμα, η 13. Λοιπόν, 5 από το σύστημα βάσης, αυτό οδηγεί σε 17,2 και στρογγυλοποιείται σε 18. Στο τέλος η Μάλτα παίρνει την βάση 5 και μισή έδρα με το διαιρέτη και καταλήγει στις 6 έδρες. Βλέπετε επίσης και την Γερμανία που είναι ο ανώτερος αριθμός και οδηγεί στο 96. Τώρα, η αναλογικότητα όμως μειούμενη προς τα κάτω. Η πρώτη στήλη υπολογίζεται χωρίς τη στρογγυλοποίηση. Η δεύτερη στήλη με την, προειδο... στρογγυλοποίηση. Η πρώτη στήλη είναι ο πληθυσμός αλλά έχει διαιρεθεί με τον διαιρέτη τον οποίο είπα και βλέπετε πώς λειτουργεί ο τύπος αυτός. Οι αριθμοί τους οποίους βλέπετε μειώνονται οι αριθμοί αυτοί όσο μειώνεται και ο αριθμός του πληθυσμού. Δεν μπορεί να παραδιαστεί αυτή η αρχή. Και μετά κάνουμε τη στρογγυλοποίηση. Η στρογγυλοποίηση οφείλουμε να την κάνουμε όπως είπα, είναι μια ανθρώπινη θα έλεγα προσπάθεια, λογική και όχι μαθηματική Και αν κοιτάξει κανείς τους αριθμούς αυτούς, αφού έχουμε εφαρμόσει λοιπόν τη στρογγυλοποίηση, θα δει ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις όπου παραβιάζεται ουσιαστικά η ερμηνεία Λαμασούρ Σεβερίν. Βλέπετε λοιπόν στην πρώτη περίπτωση αυτό ε, συμβαίνει σε περιοχές όπου υπάρχουν ομοιότητες. Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία, γύρω στα 60 εκατομμύρια. Η στρογγυλοποίηση λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που δίνει τη δυνατότητα στη Γαλλία να έχει ένα λόγο ο οποίος είναι μικρότερος όμως από ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία. Οι στρογγυλοποιημένοι αριθμοί για την Γαλλία δίνουν 79,02 έδρες. Αυτό το 79,02 μη σας κάνει εντύπωση γιατί είναι υποχρεωτικά ότι πριν γίνει η στρογγυλοποίηση θα υπάρχουν αποστάσεις από την πορεία προς τη στρογγυλοποίηση και η Πορτογαλία το ίδιο βρίσκεται και αυτή ε, πάρα πολύ κοντά, έχει 12,99, είναι πάρα πολύ κοντά στον ακέραιο αριθμό, ενώ η Γαλλία είναι πάρα πολύ μακριά. Αυτά όμως εξαρτώνται όπως είπα από τον αριθμό του πληθυσμού και αυτά μπορεί να αλλάξουν με το χρόνο. Λοιπόν, αυτές ε, οι διαφοροποιήσεις από τη μέθοδο Λαμασούρ, Σεβερίν, είναι αναπόφευκτες αν θέλετε, αν και δεν είναι ευχάριστες. Βέβαια μαθηματικοί είμαστε, μπορούμε να κάνουμε τις απαιτούμενες διορθώσεις, αλλά οι απαιτούμενες αυτές μαθηματικές διορθώσεις δεν θα είναι διαφανείς στην ανάγνωσή τους, στην πολιτική τους ανάγνωση. Είναι προτιμότερο λοιπόν να ακολουθήσουμε μία φόρμουλα η οποία να είναι εύκολα επεξηγήσιμη, ακόμα αν και στις περιπτώσεις τρογγυλοποίησης ίσως να υπάρχουν ίσονες παραβιάσεις της αρχής Σεβερίν Λαμασούρ. Τώρα, αυτά τα οποία σας είπα ήταν για 27 χώρες μέλη. Τώρα ας περάσουμε στις 28 χώρες. Προστίθεται εδώ η Κροατία, δηλαδή στην θέση 21 πληθυσμιακά. Η Κροατία θέλει 11 ένδρες. Οι έδρες αυτές από κάπου θα πρέπει να προέλθουν. Ο επόμενος πίνακας αφορά 29 χώρες. Η Ισλανδία είναι μια μικρή χώρα. Και αυτές οι έξι έδρες που θα πάρει μια τόσο μικρή χώρα και αυτές από κάπου πρέπει να βγουν. Και γι' αυτό θα ήθελα αφού σας τα παρουσίασα αυτά να πω ότι υπάρχουν ίσως κάποιοι τομείς τους οποίους θα υπάρξουν απορίες, κάποιοι τομείς τους οποίους μπορώ να δώσω κάποιες απαντήσεις Μία ερώτηση είναι σαν παράδειγμα τι θα συμβεί αν υπάρξει μία ένταξη κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής περίοδου. Αυτά είναι θέματα στα οποία εγώ σχόλια μικρά μόνο μπορώ να κάνω και μπορώ αν θέλετε να σχολιάσω σαν μαθηματικός γιατί επιλέξαμε τη στρογγυλοποίηση προς τα άνω και γιατί χρησιμοποίησαμε σαν βάση τον αριθμό 5. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά για την παρουσίαση και για την εργασία σας. Αυτά που είπατε θα πρέπει να τα χωνέψουμε θα έλεγα προσεκτικά κατά τη διάρκεια των επομένων προεκλογικών εκστρατιών. Θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα στον κύριο Ντάφ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Κρίμετ γιατί έκανε μια ιδιαίτερη προσπάθεια να μας βοηθήσει σε επίπεδο πρακτικό. Και να τον ευχαριστήσω επίσης διότι ήταν διευθύνων αυτή της ομάδας η οποία συναντήθηκε στο ΚΕΜΠ και επέδειξε ιδιαίτερες συντονιστικές ικανότητες σε αυτό το συμπόσιο. πάντα υπήρχε σαν στόχος θα έλεγα κάποιες προτάσεις τις οποίες θα μας έκαναν κάποιοι μαθηματικοί, μαθηματικοί οι οποίοι μετά από δύο μέρες συνάντησης θα κατέληγαν σε μια συμφωνία. Στο παρελθόν πάνω σε αυτό το θέμα έχουν υπάρξει αρκετές μεμονωμένες προτάσεις θυμίζω προτάσεις οι οποίες ε, χαρακτηρίζονται από ε, διφορούμενες απόψεις πολλές φορές από τους επιστήμονες σχετικά με το ποια είναι η πιο κατάλληλη λύση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν θεωρώ ότι οι συζητήσεις οι οποίες έγιναν ήταν ιδιαίτερα παραγωγικές όσο μπορούσα να τις κατανοήσω βέβαια. Μετά από όσα άκουσα η γνώση μου των μαθηματικών αυξήθηκε ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο από τότε που έφυγε από το σχολείο βέβαια και πάει πολύ καιρό. Αλλά ήταν μια συζήτηση ιδιαίτερα κακοφόρα. Και νομίζω ότι μου απέδειξε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχει μαθηματικός τύπος που να λύνει το θέμα αυτό, είναι κάτι το δυνατό. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις στην πρόταση Λαμπασούρ Σεβερίν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί όπως γνωρίζετε η πρόταση αυτή δεν έχει θα έλεγα νομιμοποιηθεί τυπικά στα πλαίσια επίσης και της πράξης του 1976. Θα ήθελα επίσης να πω ότι μου αρέσει η αντιμετώπιση βάση συν στρογγυλοποίηση. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή, όπως είπε ο καθηγητής, είναι συμβατή με τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου Και από την άλλη η πρόταση αυτή είναι συμβατή με την αρχή της δημοκρατίας η οποία λέγει ε, ένας πολίτης έχει δικαίωμα σε μία ψήφο. Θεωρώ ότι είναι σωστή επίσης και η επιλογή της τρογγυλοποίησης προς τα άνω Πρόκειται για μια απόφαση η οποία είναι πιστή. Στην αρχή της μειούμενης αναλογικότητας έτσι όπως έχει διατυπωθεί, γιατί είναι κάτι το οποίο συνολικά θα έλεγα στο τέλος ευνοεί τις μικρότερες χώρες. Να υπενθυμίσουμε εδώ γιατί εμείς σαν Επιτροπή αναζητούμε να κάνουμε μια τέτοια μαθηματική πρόταση. Πρώτον, γιατί πιστεύουμε ότι μια τέτοια πρόταση δεν μπορεί παρά να είναι δικαιότερη από την σημερινή κατανομή. Τη σημερινή κατανομή, η οποία είναι προϊόν, θα έλεγα, πολιτικού παζαρέματος ή ιδιαίτερα αδιαφανούς. Στο τέλος της διακυβερνητικής διάσκεψης όπου δεν υπάρχει τίποτα άλλο πλέον προς διαπραγμάτευση. Θεωρώ παράλληλα ότι είναι σημαντικό να είμαστε όλοι δικαιότεροι, αλλά ταυτόχρονα και να διασφαλίζουμε την απαραίτητη διαφάνεια. Και γι' αυτό η πρόταση του Cambridge σίγουρα καταφέρνει αυτά να τα συνδυάζει. Ένα τελικό σημείο. Οι έδρες οι οποίες κατανέμονται με το σημερινό καθεστώς ξεκινούν με ίση βάση για κάθε χώρα. Δηλαδή 5 και στρογγυλοποιούμενο 6 και αντιπροσωπεύουν το 25 περίπου της 100 του συνόλου των εδρών στην Ολομέλεια. Όσο προχωρούμε με τις εντάξεις νέων χωρών θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις έτσι ώστε είτε να εμείνουμε σε αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο, σε, αυτόν, σε αυτή τη σχέση αν θέλετε και αν αποφασίσουμε πολιτικά ότι κάτι τέτοιο είναι σωστό και το θεωρώ αυτό σωστό είναι απαραίτητο στο μέλλον να κατέβει η βάση από 5 σε και οι μαθηματικοί προτείνουν εδώ ότι αν είχαμε 32 χώρες μέλη σαν παράδειγμα, ίσως η βάση θα έπρεπε να κατέβει ακόμα περισσότερο και να φτάσει ίσως και σε, στο 3 αντί για το 5. Εάν λοιπόν καταλήξουμε στο να δεχτούμε την πρόταση αυτή σαν βάση διαπραγμάτευσης πλέον με το Συμβούλιο τα πράγματα δεν θα εξαρτηθούν πλήρως από εμά για να ληφθεί η απόφαση Παρ' όλα αυτά θα εξαρτηθεί από εμά να γίνει αυτή η πρόταση και να ξεκινήσουν οι συζητήσεις με το Συμβούλιο. Νομίζω ότι οι συζητήσεις αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και νομίζω ότι όπως προβλέπετε, έχουμε τις δυνατότητες να σταθεροποιήσουμε το σύστημα όσο αυξάνεται και ο αριθμός των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ακούσω και τις αντιδράσεις των συναδέλφων από πλευράς του καθηγητή Γκρίμετ. Θυμίζω βέβαια ότι ο καθηγητής Γκρίμετ θα μας δώσει την τελική του έκθεση σε λίγες εβδομάδες. Και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα εξετάσουμε αυτά λεπτομερέστερα. Και σαν εισηγητής γύρω από το θέμα αυτό, ελπίζω ότι θα έχουμε την δυνατότητα περαιτέρω συζήτησης και στην επόμενη συνάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον Άντριου Νταφ και φυσικά και τον καθηγητή Γκρίμετ για την παρουσίασή του και τα απορίσματα του συμποσίου του Κέμπριτζ. Εγώ χαιρετίζω αυτή την παρουσίαση γιατί ε, μας απαντά στα ζητούμενα που είχαμε θέσει εκτός από ένα αμφισβητούμενο επιστημονικά ζητούμενο που αφορά στην ε, αναλογικότητα, την μειούμενη αναλογικότητα στη φθήνους αναλογικότητα που φαίνεται ότι δεν είχε ιδιαίτερα ισχυρές βάσεις. Η επιλογή της μεθόδου της Fix Prop δηλαδή μία σταθερής βάσης που σέβεται την αρχή ισότητας μεταξύ των κρατών μελών και την αναλογικότητα. Επιλέξαμε λοιπόν την πιο αναλογική μέθοδο, την πιο δυνατή αναλογική μέθοδο μέσα στα πλαίσια της θύνουσας αναλογικότητας. Και αυτό τονίζεται από την επιλογή της βάσης 5 και όχι 6. Εν μέρη είναι σωστή. Με την επιλογή βέβαια του στρογγυλέματος προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Και αυτό εξισορροπεί κάπως τα πράγματα προς ε, τις μικρομεσαίες χώρες. Αυτά τα λέω ξανά εγώ, τα επαναλαμβάνω για να με διορθώσετε αν δεν κατάλαβα καλά. Λογικό μου φαίνεται όλα αυτά. Αλλά α, νομίζω το πρόβλημα θα είναι οι επιλογές ε, ε, και τα πολιτικά παραπι... ε, παρατράγουδα που θα προκύψουν γιατί επιλέξατε το 5 και όχι το 6, γιατί κάνετε αυτή την ανακατανομή έναντι μιας ιστορικής πρακτικής που μπορεί να έχει πολιτικές, ε, φανερές πολιτικές επιπτώσεις σε αυτό το κοινοβούλιο, πέρα από το Συμβούλιο δηλαδή. Όντας ε, εγώ εξ αρχής υποστηριχτής της ε, γραμμής fix prop ως λογικής γραμμής υπολογισμού, Θεωρώ ότι ο συμβιβασμός που προσεγγίσαμε είναι πάρα πολύ θετικός και ελπίζω ότι η λογική και η ορθολογική θα επικρατήσουν εδώ στο σώμα και θα μας επιτρέψουν να πρικοδοτήσουμε το Συμβούλιο με ένα διαφανές και αντικειμενικό σύστημα. Ευχαριστώ κύριε Γκουαλτιέρη. Ο κύριος Χέφνερ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο καθηγητή και τους υπόλοιπους μαθηματικούς και ιδιαίτερα τον Άνδριο Νταφ για αυτή την πρωτοβουλία. Και θεωρώ πως είναι προφανές και πως θα ήταν αλλιώς πως ε, υπάρχει μια μαθηματικά καθαρή δυνατότητα να εφαρμοστεί η αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας και μάλιστα καλύτερα από ό,τι θα γινόταν με ένα πολιτικό παζάρι. Και νομίζω πως μακροπρόθεσμα καλό θα είναι για εμάς να βρούμε ένα τέτοιο μαθηματικό τύπο ο οποίος θα είναι απλός, διάφανος και θα αποφεύγει κάθε οσμή αυθαιρεσίας. Έχω όμως κάποιες ερωτήσεις, μια που έχουμε την ευκαιρία να ευθύνουμε αυτές τις ερωτήσεις. Βεβαίως, είναι σαφές πως η χρήση του μαθηματικού τύπου θα γίνει στο πλαίσιο ενός υπάρχοντος πολιτικού πλαισίου, δηλαδή ο βασικός, η βάση του αριθμού 6, 5 συν 1, το επιλέξατε γιατί βεβαίως αντιλαμβάνεστε πως ε, και οι λαοί μας ε, το έχουν ε, ε, έτσι δεχτεί και το ίδιο για το 96 και για το 751 που είναι πολιτικά δεδομένα και λογικά. Ε, ένα δεν καταλαβαίνω. Επιλέξατε έναν διαιρέτη ο οποίος δίνει τη δυνατότητα όλες οι χώρες ε, χρησιμοποιώντας τη φθήνουσα αναλογικότητα να οδηγηθούν σε μια αναλογική εκπροσώπηση του πληθυσμού τους και είπατε πως αν πέφτουμε σε κάποιο δεκαδικό είπατε πως η στρογγυλοποίηση προς τα πάνω είναι ισχύ της μικρής χώρες κάτι που εγώ βρίσκω λογικό ένα πράγμα λοιπόν δεν καταλαβαίνω είπατε στην περίπτωση της ε, Γερμανίας δεν κάνατε στρογγυλοποίηση αλλά ε, προς τα πάνω, κάνετε ε, μια στρογγυλοποίηση προς τα κάτω. Δεν ξέρω, και δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσουμε και στο γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο. Ναι, ναι, είναι στη συνθήκη, δεν είμαι μαθηματικός, αλλά τόσα μαθηματικά και εγώ μπορώ να, το, να τα καταλάβω. Δηλαδή, εάν δεχτείτε αυτά τα δύο δεδομένα, το 6 ως κατώτατο και το 96 ως ανώτατο, μπορείτε να επιλέξετε έναν διαιρέτη που θα φτάσει στο 96 για να μην πάμε από το 105 στο 96. Εντάξει, καταλαβαίνω στρογγυλοποίηση το, το 0,1 και ξέρω εγώ 0,89 και όλα αυτά τα στρογγυλοποιείτε προς τα πάνω. Σε μία περίπτωση στρογγυλοποιείτε προς τα κάτω, την περίπτωση της Γερμανίας. Αυτό νομίζω είναι εδώ πέρα, έχει επιλεγεί αυθαίρετα και πολιτικά. Και, γιατί... Τι με ενδιαφέρει αυτό το οποίο συζητούμε εδώ πέρα να γίνει αποδεκτό και στην πατρίδα μου. Και αυτός ο τύπος μάλλον, μπορώ να σου το πω από τώρα δηλαδή, δεν θα γίνει αποδεκτός. Γι' αυτό θέλω να σας παρακαλέσω, να σας ζητήσω να μας ε, βάλετε έναν υπολογισμό που θα χρησιμοποιεί τον διαιρέτη, δηλαδή να είναι κάπως πιο μικρός, ε, κατά τρόπον ώστε να χρησιμοποιείται η ίδια αρχή για όλους. Εκεί δηλαδή που δεν υπάρχει ολόκληρη έδρα, να ακολουθήσουμε την ίδια στρογγυλοποίηση και στα 27 κρατη Για να καταλήξουμε στα 96 κανονικά και όχι σε μία μόνο περίπτωση να στρογγυλοποιήσουμε προς τα κάτω. Ε, ευχαριστώ κύριε Ο Φόξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Άντριου για την έκθεση αυτή. Θα θυμάται πω όταν συζητήσαμε στο παρελθόν εκλογικές μεταρρυθμίσεις, εγώ δεν δεν ήμουν και πάρα πολύ υπέρ, αλλά η εισαγωγή ενός μαθηματικού τύπου νομίζω είναι η πιο λογική πρόταση και ευχαριστώ τον καθηγητή τον κύριο Γκρίμετ για τις σαφείς εξηγήσεις του. Νομίζω πως ο τύπος στον οποίο κατέληξε είναι διαφανής, είναι σαφής και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να εξηγήσουμε στους ψηφοφόρους μας. Και αυτό είναι πλεονέκτημα. Και επίσης θα τελειώσει, όπως είπε και ο Άντριου, το παζάρι που εμφανίζεται σε κάθε διακυβερνητική διάσκεψη. Επίσης, αποδέχομαι αυτό το οποίο είπε ο Άντριου, πως πρέπει να δούμε το ζήτημα του αριθμού βάσης ε, στον τύπο αυτόν. Γιατί θα απαιτηθεί εδώ πέρα αλλαγή της συνθήκης και αυτό θα είναι δύσκολο. Τόσο θα επανέλθω σε αυτό. Οπότε, θεωρώ χρειάζεται ως μέρος αυτού του τύπου να πείτε κάτι που θα λέει πως ο αριθμός ο βασικός δεν θα υπερβαίνει το 20% παραδείγματος χάρη, του συνολικού αριθμού εδρών. Φτάσατε στο... Ο Άντριου λέει 25%, εγώ είπα 27,5%. Και 135 στους 751 είναι 18%. Τώρα δεν ξέρω, εάν θεωρήσουμε το 20% ως απόλυτο μάξιμου και αν φτάσουμε εκεί να μειωθεί κατά έναν, Νομίζω μπορεί να το διατυπώσει καλύτερα ο καθηγητής, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη, νομίζω, την πιθανότητα περαιτέρω εντάξεων κρατών στην Ένωση. Οπότε ο καθηγητής έκανε τη δουλειά του, κατέληξε ένα μαθηματικό τύπο και τώρα επαφίεται στου πολιτικού στη συνέχεια. Και φοβάμαι πω ε, τα σχόλια του κυρίου Χέφνερ ε, αποκαλύπτουν τη δυσκολία στο να συμφωνήσουμε σε κάποιον τύπο, γιατί αν δείτε τον πίνακα 27 θα δείτε πως 16 χώρες χάνουν ευρωβουλευτές. Εάν είστε η Πορτογαλία, από τους 22 πάτε 18. Είναι σημαντικό ποσοστό των ευρωβουλευτών. Και βεβαίω απαιτεί ο τύπο αυτός ομοφωνία. Και εδώ πέρα αντιλαμβάνομαι το δύσκολο έργο του Άντριου που πρέπει να πείσει 27 κρατημέλη πως είναι καλή αυτή η ιδέα. Όταν 16 από αυτά θα χάσουν Έδρε. 6 μόνο θα κερδίσουν και ένας λόγος για τον οποίο είναι υπέρ είναι πως το Ηνωμένο Βασίλειο κερδίζει έξι έδρες. Οπότε η δική μου η περιφέρεια, τα νοτιοδυτικά, θα πάνε από τις 6 σε 7 και εγώ θα βγω ευκολότερα. Αλλά θεωρώ πως η πολιτική πτυχή θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και αν μπορώ να το θέσω ως το γερμανικό ζήτημα. Γιατί να έχει πλαφών 96 Γερμανία. Η απάντηση είναι για το γράφει η συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά εάν είναι να πούμε πως θα ξαναγράψουμε τον τύπο, τότε σωστά θα ρωτήσει η Γερμανία γιατί να ξαναγράψουμε τα πάντα εκτός από αυτό το πλαφόν. Δεν είμαι σίγουρος πως υπάρχει λογική εξήγηση για να μείνει η Γερμανία στους 96. Είναι βολικό άμα είσαι από άλλη χώρα βεβαίως αλλά δεν είμαι σίγουρος πως υπάρχει λογικό επιχείρημα για το, για το πλαφόν της Γερμανίας 96. Ενδιαφέρουσα λοιπόν αυτή η παρουσίαση και είναι πράγματι διαφανές και σαφές το σύστημα, αλλά η πιθανότητα να συμφωνηθεί σε διακυβερνητική διάσκεψη είναι τίνουν προς το μηδέν θα έλεγα. Ο συνάδελφος Ταρκόφσκι. Uh, Ευχαριστώ κύριε καθηγητά για την σαφή σας παρουσίαση. Συμμετείχα στις συζητήσεις κάποιες κατάλαβα και σας συγχαίρω γιατί καταλήξατε σε, μια, σε έναν διαφανή τύπο και τα εξηγήσετε με έναν απλό και συνοπτικό τρόπο που δεν ήταν εύκολο. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα πολλοί δεν ξέρουν πως υπήρχε ένα σύστημα το οποίο συμφωνήθηκε σύνοδο της Κοπενχάγης και είχαμε αυτές τις δόσεις με βάση τις οποίες κατανεμήθηκαν οι έδρες. Οπότε βασιστήκαμε σε κάποιον τύπο, αλλά προφανώς μετά την αποδοχή αυτού του τύπου, μετά τα πάντα α, επαφίενται στο παζάρι μεταξύ κρατών μελών. Όταν μιλάμε τώρα, για, το περάσουμε στις λεπτομέρειες, η ιδέα του να περάσουμε στην τρογγυλοποίηση όπως την προτείνετε εσείς και η βάση είναι σωστή. Και πράγματι γιατί η βάση ευνοεί τα μεγάλα κράτη, η τρογγυλοποίηση τα μικρά, υπάρχει μια λογική. Συμφωνώ όμως πως εάν το προτείνουμε αυτό κάπου παραπέρα πρέπει να ε, αιτιολογήσουμε καλύτερα την βάση, αυτό το 6. Και είπαμε στις συζητήσεις μας πως τουλάχιστον αποδεχόμαστε αυτή τη φάση τη χαμηλότερη που θα φτάσουμε στο 6 δηλαδή. Κάπως πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό για να το καταλάβουν και οι άνθρωποι γιατί επιλέχθηκε αυτός ο αριθμός. Και μετά να πούμε ότι ούτως ή άλλως όλοι έχουν 6 έδρες και κατανέμονται μετά οι έδρες ε, ρεαλιστικά. Προφανώς το σκεπτικό εδώ πέρα της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου είναι το εάν μπορούμε να στηρίξουμε μια τέτοια θέση ή όχι και όταν ακούμε για το παζάρι που λαμβάνει η χώρα στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια για τον αριθμό των εδρών ε, ως εάν να μην ε, ήταν δυνατή η λήψη αποφάσεων ε, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ έτσι αξιοπρεπής τρόπος για την κατανομή των εδρών, αλλά απ' την άλλη πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα. Οπότε συμφωνώ πως είναι πολύ κομψός αυτός ο τύπος και σε έναν ιδανικό κόσμο η οθέτησή του θα μας επέτρεπε να δικαιολογήσουμε καλύτερα την κατανομή των εδρών. Αλλά ακόμα και από την προκαταρκτική αυτή συζήτηση βλέπουμε πως όλοι ε, δρούν εδώ πέρα υπό την εθνική τους ιδιότητα όταν το συζητάμε. Και αν δείτε το πώς έχουμε προχωρήσει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ειδικά εδώ μέσα προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα εθνικά όρια και σκεφτόμαστε στο πλαίσιο έτσι, της ευρωπαϊκής οικογένειας αλλά όταν μιλάμε για τον αριθμό των εδρών, τον αριθμό ψήφων ή τα χρήματα μια φορά βεβαίω μιλάμε ξανά με εθνική ιδιότητα και θα είναι δύσκολο αλλά ακόμα και αν αποτύχουμε, τουλάχιστον αν προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε εδώ πέρα ένα τέτοιο σκεπτικό, θα μας ωφελούσε πάρα πολύ, γιατί είναι λογικό και συνεπές. Αυτά και εύχομαι καλή τύχη. Είναι κόλπο βλέπω των ε, μαθηματικών του Κέμπριτζ να αποκτήσει η Μεγάλη Βρετανία 8 παραπάνω έδρες ε, για να μην ε, καταψηφίσουν σε δημοψήφισμα. Τέλος να περάσω να περάσω τώρα σε σοβαρές παρατηρήσεις. Εγώ προσωπικά θα το προσπέγραφα αμέσως τώρα. Είναι μια μαθηματική μέθοδος, είναι σωστό και έτσι έχουμε τους τρεις πολιτικά καθορισμένους αριθμούς 96, το 6 και το 751 και στο πλαίσιο αυτό βρίσκουμε μια λύση η οποία είναι μόνιμη και δεν χρειάζεται συνεχώς παζάρια σε κάθε διεύρυνση υπάρχει ένας μαθηματικός αυτοματισμός. Και επειδή δεν ήμουν και τόσο καλό στα μαθηματικά στο σχολείο, τόσο μπόρεσα να τα παρακολουθήσω ε, και όσο μπόρεσα ήταν ε, λογικά ως προσέγγιση. Θα ήθελα βεβαίως και τη βοήθειά σας εάν είναι να τα εξηγήσουμε. Ο κύριος Χέφνερ ανέφερε κάτι το σημαντικό. Εντάξει, οι 96 γερμανικές έδρε αναφέρονται στην συνθήκη, αλλά έχουμε πάντα στη Γερμανία τη συζήτηση το πώς μπορούμε να κάνουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία όταν δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια βασική αρχή ένα άτομο, μία ψήφος. Αρχή της δημοκρατίας. Οπότε θα θέλαμε να μας βοηθήσετε για να μπορέσουμε να αιτιολογήσουμε και πολιτικά αυτό τον αριθμό το 96 δεύτερον, για το οποίο αναφέρθηκε ήδη, πως για να περάσει κάτι τέτοιο είναι πάντα δύσκολο όταν έχουμε μία λογική λύση να περάσουμε παρόλα αυτά το ότι έχουμε μείωση για 18 χώρες. Γιατί ξέρετε εκεί πέρα σταματάει η λογική στους πολιτικούς όταν μιλάμε για μείωση. Και εδώ πέρα βλέπω πολιτικό πρόβλημα του πώς θα περάσει κάτι τέτοιο. Και ακριβώς επειδή είμαστε κάπου στις μέσες χώρες όσον αφορά την τάξη μεγέθους, θα πρέπει να γίνουν κάποιες σημαντικές εξηγήσει για να μπορέσουν να εξηγήσουν οι συνάδελφοι το πώς χάνουν αυτές τις, ε, τις έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί πέρα θα θέλαμε να μας βοηθήσετε σε κάποια άλλη ευκαιρία για με πιθανόν κάποια επιχειρήματα, κάποιες πληροφορίες για να μην ε, δράσουν και παράλογα οι ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ κύριε Μπρόκ. Κύριε Σεφ, Σεφλιν και μετά Γκρούτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρέμετ. Νομίζω ότι κάπως κατάλαβα, κάτι κατάλαβα από αυτά τα οποία είπατε. Νομίζω ότι για ανθρώπους που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα κάτι καταλάβαμε. Ίσως ένα μικρό ε, βίντεο ή ένα DVD σε 23 γλώσσες Νομίζω ότι ένα DVD λοιπόν θα δώσει περισσότερες εξηγήσει για την ανακατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που κάτι ε, τέτοιο θα ε, προσφέρει. Νομίζω λοιπόν ότι η κατεύθυνση είναι γενικά η σωστή. Η κατανομή των εδρών κατά κάποιο τρόπο καθίσταται απρόσωπη και διαφανής. Αυτό είναι αληθές. Εκεί όμως που έχω κάποιες αμφιβολίες και εδώ θα συμφωνήσω με τους κυρίους Χέφνε, Φόξ και τα λοιπά, υπάρχουν κάποια πολιτικά προβλήματα με την κατανομή. Το βλέπω και το λέω λίγο χονδρικά τώρα, αλλά τίνω να δω ότι οι μεσαίες χώρες φαίνεται ότι στριμώχνονται, ακόμα και η δική μου, η Ουγγαρία από 22 πηγαίνουν σε 18. Αυτό είναι κάτι που δεν θα περάσει εύκολα. Και δεν θα μας αρέσει κάτι τέτοιο. Και ιδιαίτερα οι μεγάλες χώρες φαίνεται ότι πηγαίνουν μια χαρά. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, ε, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ρουμανία ωφελούνται από την ανακατανομή. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι σε ένα όργανο σαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ποσοστό σταθερότητας παρέχεται με το σύστημα το οποίο ουσιαστικά έχουμε κληρονομήσει. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία υπερεκπροσώπηση των μικρών κρατών, είτε μας αρέσει είτε όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο στην ουσία θα έλεγα κρατάει και την ισορροπία ανάμεσα στη Σκοτία, την Ουαλία και, το, και, και την Αγγλία γενικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό δεν είναι ο δικός σας στόχος. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας να προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε με τέτοιο τρόπο γιατί οι Ούγγροι δεν θα συμφωνήσουν με μια τέτοια πρόταση και εγώ θα ακούσω επιχειρήματα και όσο έξυπνος και αν θεωρώ ότι είμαι δεν θα εξηγήσω το πώς θα πέσουμε από 22 σε 18. Ήδη ήμασταν 24 και πήγαμε 22, μετά θα πάμε 18 και μετά θα πάμε 15 και τι γίνεται από εκεί και πέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τα επιχειρήματα τα οποία θα ακουστούν στο μέλλον. Εύνερ, Α, όχι, όχι, λάθος. Ευχαριστώ κύριε Κασίνη. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Κρίμετ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η πρόταση την οποία κάνετε. Αυτό το οποίο μου δημιουργεί πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η στρογγυλοποίηση. Αν το εξηγήσω αυτό σε ένα μαθηματικό ή σε ένα έμπορο, το θέμα της στρογγυλοποίησης στην ουσία είναι κάτι το πάρα πολύ συγκεκριμένο ενώ εμείς εδώ βλέπω ότι στρογγυλοποιούμε συστηματικά προς τα πάνω. Θυμίζω επίσης ότι το 90% των βουλευτών δεν είναι μαθηματικοί. Εγώ μηχανικός είμαι, αλλά δεν σας κατανοώ απόλυτα παρά την πανεπιστημιακή μου κατάρτιση. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα εδώ με τους αριθμούς και οι αριθμοί ε, νομίζω πρέπει να παρουσιαστούν με πιο ξεκάθαρο τρόπο σε περίπτωση της διεύρυνσης. Όπως είπε και ο κύριος Μπροκ και οι άλλοι, το θέμα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι θέμα επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι δύσκολο πράγμα. Όλοι οι ευρωσκεπτικιστές στη χώρα μου θα χειροκροτήσουν ε, όταν παρουσιαστεί η μαθηματική αυτή πρόταση η οποία θα τροφοδοτήσει είναι σαφές τα επιχειρήματά τους κατά της Ευρώπης. Νομίζω ότι θα, βρεθεί, θα πρέπει να βρεθεί προς τα πάνω και προς τα κάτω ένας διαφορετικός τρόπος στρογγυλοποίησης. Υπάρχουν ε, πολιτικά κριτήρια τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν αν δεν μεσολαβήσει μια νέα συνέλευση, κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. Είναι σαφές λοιπόν ότι ο τρόπος στρογγυλοποίησης προς τα άνω και προς τα κάτω είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Δεν ξέρω, μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε καλύτερα το πώς προχωράτε στη στρογγυλοποίηση. Κατανοώ για τις μικρές χώρες ότι θα πρέπει να υπάρξει στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, αλλά γιατί ε, να μην παρουσιάσουμε με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα, πιο απλό τρόπο, πιο επεξηγήσιμο, έτσι ώστε στις εκλογικές μας περιφέρειες να καταλάβουν και οι απλοί άνθρωποι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέφνερ, ναι, ζήτησα ξανά τον λόγο για πριν απαντήσει ο κύριος καθηγητής γιατί κατάλαβα νομίζω πως υπήρχε μια παρανόηση εδώ πέρα το ζήτημα δεν είναι τα εθνικά συμφέροντα απλά επειδή εδώ πέρα ακολουθούμε μια μαθηματική μέθοδο. Απλά αναρωτιέμαι γιατί εγώ πρέπει συνέχεια να αγωνίζομαι να εξηγώ στους ε, ψηφοφόρους μου πως εδώ λειτουργούμε με βάση την αρχή ένα άτομο μία ψήφος αλλά αυτό και γιατί αυτό είναι θετικό το ότι δηλαδή έχουμε αναλογικά πάντα λιγότερους βουλευτές από την ε, Μάλτα. Οπότε καλό θα ήταν να βρούμε έναν τύπο ο οποίος θα μπορεί να εξηγήσει κάτι τέτοιο. Δεύτερον, συμφωνώ πλήρως με τα πολιτικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν ε, ως προϋποθέσεις, δηλαδή το 6 ως βάση, το 96 ως πλαφόν, το 751 ως σύνολο. Και τον τύπο τον οποίον ε, βρήκατε να σας πω πώς το βλέπω εγώ δηλαδή. Έχετε ένα διαιρέτη, αναζητήσατε έναν διαιρέτη ο οποίος εντό αυτού του πλαισίου οδηγεί σε μια α, φθήνουσα αναλογική κατανομή. Ένα ξεκάθαρο πράγμα δηλαδή και δεύτερον εκεί πέρα όπου είχαμε μία κέραιος, όπου είχαμε δεκαδικούς κατά κανόνα δηλαδή, εφαρμόσατε τον κανόνα στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω. Ναι, συμφωνώ, αλλά το συζητάμε αυτό, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου. Αυτό το οποίο έχει πολιτικές συνέπειες πρέπει να το συζητάμε πολιτικά. αλλά εμένα το θέμα μου αφορά αυτή τη στιγμή αποκλειστικά τα μαθηματικά. Και θέλω να, το πω ξεκάθαρα. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ε, παίρνετε το 6 και το 96 κάτω έχετε το, τις 300.000 Μάλτας και πάνω τα 82 εκατομμύρια της ε, Γερμανίας και γιατί δεν υπολογίζεται άρα έναν διαιρέτη να ε, ισχύει για όλους. Σας το λέω, είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις με την απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού ε, Δικαστηρίου και θα μπορέσουμε να το αντικρούσουμε αυτό πολιτικά εάν πούμε πως εδώ πέρα δεν υπάρχει αυθαιρεσία. Και να πούμε πως βρήκαμε ένα συντελεστή ο οποίο ισχύει για όλου. Δηλαδή, εγώ τι θα του πω, έχουμε ένα συντελεστή που ισχύει για 26 χώρε και μόνο για τη Γερμανία, όχι. Θα ήθελα δηλαδή ε, να μου πείτε ποια, γιατί σε αυτή τη μία περίπτωση κρίνατε πολιτικά και στι υπόλοιπε ακολουθήσατε ένα μαθηματικό τύπο θα μπορούσαμε να έχουμε, αν θέλετε, ένα υπόδειγμα, έναν τύπο, ο οποίο θα ενισχύει πράγματι ναι, τι μικρέ χώρε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά εδώ πέρα ο τύπο δεν ισχύει για όλου. Αυτό είναι, αυτή είναι η δυσκολία μου. Α, Ταρκόσκι, Κύριο Ταρκόσκι. Να δώσω μία εξήγηση, ε, Γκέραρτ γιατί είπε ε, πως παρεξηγήσαμε όταν είπα εγώ πω μιλάμε υπό την εθνική ιδιότητα. Ε, δεν σημαίνει πως θέλουμε να υπερασπίσουμε εθνικά συμφέροντα, αλλά σκεφτόμαστε σε εθνικό πλαίσιο όταν λέμε πως, το πώ θα τεκμηριώσουμε τη θέση μας. Και μια που γίνεται αυτή η συζήτηση, να σα πω και άλλη μια δυσκολία. Η δυσκολία με αυτό το σύστημα είναι πω συνήθω όταν διαπραγματευόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα είναι πακέτο, γιατί διαπραγματευόμαστε διαφορετικά συστήματα. Και παραδείγματο χάρη στην περίπτωση τη Γερμανία, όταν το διαπραγματευτήκαμε αυτό μαζί με τον αριθμό των ψήφων στο Συμβούλιο, μπορεί να τεκμηριωθεί έτσι ευκολότερα η γερμανική θέση, γιατί είπαμε πως ήταν μια συμφωνία πακέτο έχουμε νέο σύστημα διπλής πλειοψηφίας και κερδίζει έτσι η Γερμανία ως πιο πολυπληθής και άρα συμφωνήσαμε να περιοριστεί ο αριθμός των Ευρωβουλευτών σε 96. Οπότε όταν εξηγήσει κανείς το πακέτο, τη λύση πακέτο, εξηγούμε καλύτερα τη θέση μας. Αλλά βεβαίως μετά πάμε αλλού, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να σκεφτούμε ξεκάθαρα με βάση ένα μαθηματικό τύπο ενώ διαφορετικά, 5-6 διαφορετικά ζητήματα. Αυτό είναι πολιτικά δύσκολο. Αλλά όταν α, ε, κοιτάξαμε το μαθηματικό τύπο δεν, δεν υπήρχε άλλη διέξοδος. Νομίζω λοιπόν αυτό είναι το πιο βιώσιμο που μπορούσαμε να έχουμε, αλλά έχουμε και τα δεδομένα πολιτικά προβλήματα. Και αυτό είναι φυσικό, ε, ειδικά να το συζητήσουμε ασύνδετα με το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Και αυτή είναι η βασική δυσκολία, γιατί πάντα υπάρχει ένα πακέτο. Δηλαδή κάποιος παίρνει έναν επίτροπο, κάποιος παίρνει ψήφους στο Συμβούλιο και μετά συμφωνούμε στι έδρε. Αλλά από τη δική μας σταθήση αυτό είναι το δίλημα που πρέπει να λύσουμε εμείς ως βουλευτές. Και εντάξει, ίσως υπερβάλλω λίγο εδώ πέρα. Ήταν και λίγο υποτιμητικό να ακούει κανεί. ε, ε σκάστε τώρα, εν πάση περιπτώσει πήρατε και δύο έδρε παραπάνω στο, στο κοινοβούλιο αλλά πολιτικά ε, όλοι συμφωνούμε πως είναι πάρα πολύ δύσκολο ειδικά για τις χώρες που χάνουν και για να πούμε την αλήθεια προφανώς ακόμα και αν σκεφτούμε το σύστημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κτλ και εγώ κοιτάω πόσες έδρες έχει η Πολωνία όχι για εθνικού συμφέροντος αλλά για να μιλήσω στους ψηφοφόρου μου είναι φυσικό Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον καθηγητή Γκρίμιτ. Πριν του δώσω το λόγο, θα ήθελα και εγώ να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Είδατε ότι κατά τη διάρκεια της συζήτηση εγώ έγραφα, έκανα πράξεις, δεν έχω υπολογιστεί μαζί μου βέβαια και έχω κάνει πάρα πολλά λάθη, φοβάμαι. Άκουσα τα κριτήρια τα οποία ακολουθήσατε και πάνω σε αυτά θα ήθελα τη γνώμη σα. Αν κατάλαβα καλά, η Γερμανία και οι χώρες από την άλλη που έχουν μόνο έξι βουλευτές και αν δεν προστατευθούν από τη συνθήκη δεν θα έχουν τον ελάχιστο αριθμό ευρωβουλευτών. Στην ουσία είναι εκτός κανόνα. Αλλά οι χώρες που είναι ακριβώς πέραν του ανωτάτου ορίου και του ελαχίστου ορίου θα πρέπει να συζητηθεί με διαφορετικό τρόπο. Μία χώρα ας πούμε με 10 εκατομμύρια και μία χώρα με 60 εκατομμύρια δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Γιατί ακριβώς αυτή που έχει 60 εκατομμύρια, ακόμα και αναφερθεί η βάση, έχουν έξι, έχει 6 φορές περισσότερα ε, πληθυσμό από τη χώρα που έχει 10 εκατομμύρια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει ακρίβεια στους υπολογισμούς και με βάση τους δικούς μου υπολογισμούς αν και επαναλαμβάνω ίσως έχω κάνει πολλά λάθη μου δίνουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πιο κοντά σε αυτά τα οποία έχουν προταθεί σύμφωνα πάντα με βάση το 6 και όχι με βάση το 5. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας το ανώτατα και τα κατώτατα όρια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αναλογικότητα ανάμεσα στις ενδιάμεσες χώρες, μικρές ή μεγάλες. Αυτό σαν σκέψη είναι σωστό ή όχι. Δεύτερον, δεν κατάλαβα καλά, και αυτό μάλλον είναι δικό μου λάθος, δεν κατάλαβα καλά γιατί επιλέξατε το 5 και όχι το 6, που θα ήταν το ελάχιστο το οποίο ουσιαστικά προβλέπετε από τη συνθήκη. Τρίτον, Είμαστε σίγουροι ότι αυτού του τύπου οι υπολογισμοί τους οποίους προτείνεται λαμβάνουν υπόψη τους ακόμα και μια μελλοντική διεύρυνση της Ένωσης προς χώρες οι οποίες είναι αρκετά μικρές. Ε, Ισλανδία, Κροατία βέβαια. Η λογική αυτή όμως θα ισχύσει αν μπουν και χώρες με πληθυσμούς μεγαλύτερους με αυτούς της Γερμανίας και αναφέρομαι στην Τουρκία. Νομίζω ότι έχετε εδώ αρκετό υλικό για να απαντήσετε. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τέθηκαν πολλές ερωτήσεις. Δεν, ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος ότι τις κατάλαβα όλες. Yeah. Ε, θα απαντήσω τέλος πάντων. Θα μείνω στην ειδικότητά μου. Το ένα είναι το 696 και το 751 και τι μπορούμε να κάνουμε. Το μεγαλύτερο κράτος θεωρείται πως, δυσ... θεωρεί πως δύσκολα θα εξηγήσει αυτό το πλαφόν. Βεβαίως το πλαφόν το μέσα στα νούμερα που μας είχαν δώσει. Και αν έχουμε το μικρότερο κράτος με 6 και το μεγαλύτερο με 96 και υιοθετήσουμε την αναλογικότητα στο ενδιάμεσο, ε, κάπου πρέπει να, να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει είναι το μέγεθος του Κοινοβουλίου, το 751. Αλλιώς μπορούμε να τραβήξουμε μια ευθεία γραμμή από το 6 έως το 96 με βάση τον πληθυσμό, αλλά δεν το έκανα γιατί θα έχαναν περισσότερα από 16 κράτη-μέλη. Γιατί έτσι θα μειώναμε αρκετά τον συνολικό αριθμό ευρωβουλευτών. Ένας άλλος τρόπος μεταξύ 6 και 96 με το μέγεθος στο συνολικό στα 751 είναι μια καμπύλη η οποία δεν θα είναι ευθεία γραμμή. Δεν χρειάζεται βεβαίως να είναι κανείς καθηγητής μαθηματικών για να, κάνει, να χαράξει μια καμπύλη. Βάζουμε τα νούμερα στο Excel και φτιάχνει μια καμπύλη μόνο του. Μετά συναντάμε κάποιον άντρα γυναίκα στον δρόμο και λένε πώς το κάνατε. Και λέμε, α, έβαλα τα νούμερα στο Excel. Δεν πιστεύω πως είναι λογικός τρόπος κατανομής εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτός, με βάση κάποια αρχή. Και αν δημοσιοποιηθεί αυτή η μέθοδος, μπορεί ο κόσμος να αμφισβητήσει την δικαιοσύνη αυτής της κατανομής. Ναι, αλλά θέλω να είμαι προσεκτικό σε πάση περιπτώσει, να μην βγω εκτό εντολή. μου. Είμαι μαθηματικός, αλλά είμαι και άνθρωπο. Εάν μας δώσουν άλλους κανόνες, εάν μας πούνε παραδείγματο χάρη πως η χώρα του αντιπροέδρου, τον οποίο τυχαίνει να ξέρουμε πρέπει να έχει ένα αριθμό εδρών, τότε μπορούμε να σκεφτούμε αυτούς τους κανόνες και να βρούμε κάποιες μεθόδους με βάση αρχές για να τηρήσουμε και αυτόν τον κανόνα, αλλά δεν μας είπαν αυτό. Λοιπόν, είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση γιατί θέτει σε εσά το ερώτημα του τι είδους κοινοβούλιο, σε τι είδους κοινοβούλιο θέλετε να είστε βουλευτές. Και πώς θα το δικαιολογήσετε αυτό στους ψηφοφόρους σας και ίσως στους ψηφοφόρους των γειτονικών χωρών, όχι μόνο στη δική σας χώρα. Υπάρχουν επίσης ε, κάποιες άλλες πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Για να δω τι σημείωση κράτησα. Το ένα είναι η βάση, πώς θα αλλάξει ε, η βάση. Πρώτα απ' όλα η βάση. Θα ήθελα εδώ πέρα να βάλω μια νέα λέξη, να το πούμε minimum. Η βάση είναι αριθμός στους, ε, υπολογισμού. Το μίνιμουμ είναι ο αριθμό που λένε στην επιτροπή σα. Εμά μα είπαν 6, αδιαπραγμάτευτο 6. Μα είπαν 6 θα είναι. Η βάση είναι ο αριθμό που βάζουμε εμεί ε, ε, στον υπολογισμό για να έχουμε ένα 6 εγγυημένο. Εάν η βάση τώρα εξαρτάται από τον αριθμό κρατών μελών και τον πληθυσμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Στην Επιτροπή μου ε, είναι, ήταν σαφές πως θα έπρεπε να εξαρτάται κάτι τέτοιο γιατί επειδή είμαστε άνθρωποι με αρχές είδαμε πως υπάρχουν κάποιες πιθανές διευρύνσεις που θα καταστήσουν το μίνιμουμ ε, 6 να μην μοιάζει λογικό. Αλλά δεν ήταν εντολή μας ε, να το εξετάσουμε αυτό. Ανεξαρτήτως αυτού το συζητήσαμε είπε ώρα. Και θα υπάρξει τμήμα στην έκθεσή μας, το οποίο είναι προαιρετικό, δεν θα είναι στις εξετάσεις, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τηρήσουμε αυτές τις ε, αρχές και επαφίεται μετά στα μέλη της Επιτροπής σας να το συζητήσετε και να προτείνετε ίσως κάτι το οποίο θεωρείται ελκυστικό. Μία δυνατότητα είναι να εξετάσουμε τη... το συνολικό ποσοστό του Κοινοβουλίου που πάει στο, στο το εγγυημένο εάν θέλετε, και αν αυτό το ποσοστό θα πρέπει να έχει ένα ανώτατο όριο, αν θα πρέπει να υπάρχουν κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ. Νομίζουμε λοιπόν πως αυτή μπορεί να είναι μια πιθανή πορεία για την Επιτροπή σας και μπορούμε ξέρω, εμείς ως απλοί πολίτες να προτείνουμε κάτι τέτοιο στην Επιτροπή αλλά δεν αποτελεί μέρος εντολής μας. Να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα. Για εμάς ποιος ως βαθματική θα ήταν πιο βολικό, αλλά βεβαίω μπορεί να ήταν θέμα διαφάνειας, εάν για μαθηματικούς λόγους θα μπορούσαμε να έχουμε μια βάση η οποία δεν θα ήταν ακέραιος αριθμός. Συζητήσαμε περί και αρκετή ώρα τα πλεονεκτήματα του 5,5. Βεβαίω μετά θα ακολουθεί η στρογγυλοποίηση, αλλά θα μας επέτρεπε αρκετή ελευθερία εάν θα μπορούσαμε να συστήσουμε έναν τύπο Βέβαια εντάξει το μίνιμουμ προφανώς θα ήταν ε, ο λόγος αριθμό, αλλά η βάση θα ήταν δεκαδικός. Ε, οπότε δεν είναι μέρος της κύρια έκθεσή μας αλλά θα συζητηθεί όπως σας είπα στο τέλος της έκθεσης ω ύλη για ανάγνωση. Μια που συζητάμε τη βάση προέκυψε το ερώτημα το γιατί δεν πήραμε το 6 ως βάση. Δυστυχώς ε, έφυγε η οθόνη και άναψαν τα φώτα, οπότε δεν μπορώ να σας δείξω τη σελίδα την οποία είχα προετοιμάσει. Ε, ανταυτού, να σας πω τι έλεγε. Τα δύο συστήματα τα οποία συζητήσαμε επί μακρόν, τόσο ναι δεν μπορούμε να τα δούμε ούτως ή τα δύο λοιπόν αυτά συστήματα, το 5 συν δηλαδή που είναι η σύστασή μας και το 6 ως βάση, συν κανονική στρομπιλοποίηση, δηλαδή προς τον πλησιέστερο ακέραιο, το 6,4 πάει στο 6, 6,6 πάει στο 7. Γνωρίζαμε και το γεγονός πως το 6 είναι ο ελάχιστος αριθμός εδρών ανακράτος μέλος και μας είπαν πως πρέπει να αντιληφθούμε πως το 7 δεν είναι ελάχιστος αριθμός. Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει ε, στον πάτο μεταξύ αυτών των δύο μεθόδων κατανομής. 5 συν προς τα πάνω είναι στον πίνακα 27. Δίνει λοιπόν 6 στα τρία κρατημέλη, Μάλτα, Λουξεμβούργο και Κύπρο και 7 στο μεγαλύτερο κράτος που είναι η Εστονία. Η τωρινή κατανομή λοιπόν αυτών των κρατών μελών είναι 6 για όλους. Οπότε το αποτέλεσμα είναι πω η Εστονία θα κερδίσει μια έδρα, Άλλε χώρε ε, μένουν στα ίδια. Εάν έχουμε το 6 έστερο, τότε βεβαίω δίνουμε περισσότερα στον, σε αυτούς που είναι πιο κοντά στον πάτο. Οπότε η Μάλτα παραμένει στι 6 το Λουξεμβούργο και η Κύπρος πάνε στις 7 και η Εστονία 8. Ίσως βεβαίως αυτό μπορεί να γίνει δεκτό. Αλλά σκεφτούμε μια ελαφρά παραλλαγή στην οποία η Μάλτα κερδίζει ε, άλλους, έχει άλλους 8.000 κατοίκους Οπότε έχει αυτή τη στιγμή 412.000, βλέπετε. Αν η Μάλτα... Δεν φταίει η Μάλτα δηλαδή, με συγχωρείτε. Εάν το μικρότερο αυτό κράτος μέλος άξανε τον πληθυσμό και έφτανε στις 420.000, έχουμε μια μικρή λοιπόν αλλαγή του αριθμού του πληθυσμού και σύμφωνα με το 6 συν πλησιέστερο θα έφτανε και αυτή στις 7 έδρες αντί για 6. Και το ε, εξετάσαμε, ίσως λάθος μπορείτε να πείτε και μπορείτε να μας διορθώσετε, θεωρήσαμε πως μπορεί να πει κάποιος πως αυτό δεν τηρεί τις προϋποθέσεις για το κατώτατο όριο. Γι' αυτό πήγαμε 5 συν αντί για 6 συν. Μετά υπάρχει ένα άλλο σύστημα το οποίο θα ικανοποιήσει τους πάντες. Όχι, μάλλον όχι τίποτα δεν ικανοποιεί τους πάντες ετέθη το ερώτημα και βεβαίω δεν έχω απάντηση, αλλά μπορώ να σου πω τι θα συνέβαινε. Το γιατί το μεγαλύτερο κράτο μέλο έχει πλαφόν. Ανεξάρτητο του ποιο είναι το μεγαλύτερο κράτο μέλο και πώ μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, γιατί παρά το ότι είναι φθήνουσα αναλογικότητα, ε, παρά είναι φθήνουσα στην κορυφή. Και δεν αρέσει αυτό στου μαθηματικού, γιατί όταν έχουμε μία καμπύλη, η καμπύλη στην άκρη πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλη κλίση για αυτό το maximum πρέπει να είναι μη διαφοροποιήσιμα. Έχει γωνία. Έχει μια γωνία λοιπόν και δεν μας αρέσει. Εμάς μας αρέσουν οι ομαλές ε, καμπύλες. Οπότε ως μαθηματικοί θα ήμασταν ικανοποιημένοι να προτείνουμε κάτι το ομαλό. Εάν... Ε, σας ξήγησα λοιπόν γιατί δεν μπορούμε να πάμε από το 696 χωρίς να αλλάξει κάτι άλλο. Οπότε αν δεν αλλάξει κάτι άλλο Εάν δεν αλλάξει δηλαδή η αναλογική κατανομή των εδρών, τότε το πλαφόν του μεγαλύτερου κράτους μπορεί να έρθει. τι συνέπειε θα έχει αυτό. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κράτο μέλο έχει 96, αλλιώς θα ελάμβανε 105 έδρε. Ε, τι να γίνει θα, θα χτίσετε νέο κτίριο και εάν ε, κάθε κράτος μέλος ε, επιμείνει σε περισσότερα, τότε χτίστε ένα πολύ μεγάλο κτίριο και όλοι θα είναι ικανοποιημένοι. Αλλά βεβαίως αν, ανέβει, αν έχει περισσότερες έδρες ένα κράτος θα έχουν όλα. Τώρα βεβαίως απομακρύνομαι λίγο από τα μαθηματικά, οπότε καλό θα είναι να σταματήσω. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως ο πληθυσμός αλλάζει, ε, τα νούμερα αυτά βασίζονται στον σημερινό πληθυσμό οι πληθυσμοί αλλάζουν, οι άνθρωποι μετακομίζουν, αλλάζει η καταμέτρηση, μετριούνται καλύτερα οι πληθυσμοί. Αυτά τα πράγματα αλλάζουν, οπότε οι κατανομές αυτές είναι προσωρινές. Νομίζω λοιπόν κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν απάντησα όλες τις ερωτήσεις σας. Ευχαρίστω να, να προσπαθήσω, αλλά φοβάμαι πως ε, παρήψα δική σας ερώτηση και δεν θα το ήθελα αυτό. Οπότε να σας ξαναδώσω τον λόγο. Eh, όχι, όχι, ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πρέπει σίγουρα να το σκεφτούμε ξανά το θέμα. Σε όλα απαντήσατε, αλλά ο κύριος Ντάφ θέλει και πάλι το λόγο. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο. Δεύτερον, κάθε συζήτηση για τις εκλογικές διαδικασίες και για την ανακατανομή των εδρών γίνεται γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει ένα μόνο ιδανικό σύστημα. Ό,τι κάνουμε λοιπόν είναι στην ουσία συμβιβαστικές προτάσεις. Η αρχή της μειούμενης ή αναλογικότητας που υπάρχει στη συνθήκη είναι μία αρχή ομοσπονδιακού χαρακτήρα η οποία προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντα των μικρών απέναντι στους μεγάλους. Κάποιοι θα πούνε ότι ίσως να μην χρειαζόμαστε μια τέτοια προστασία. Αυτή όμως δεν είναι η άποψη αυτών που ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτών που συνέταξαν τη συνθήκη, μεταξύ των οποίων και το Κοινοβούλιο. Θυμίζω ότι το Κοινοβούλιο είναι σε εισαγωγικά συνένοχο στα πλαίσια της σύνταξης της συνθήκης. Αν αλλάξουμε την άποψή μας πάνω σε κάτι το τόσο θεμελιώδες είναι σαφές ότι θα πρέπει να δώσουμε πολλές εξηγήσει. Ο Ραφαέλ είπε κάτι το οποίο ήθελα να πω και εγώ, ότι η κατανομή εδρών ανακράτως στο σώμα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της απόφασης του Συμβουλίου και σε σχέση με κάτι το οποίο είναι πλέον τμήμα της συνθήκης της Λισαβόνας, κάτι το οποίο πολλοί από εμά δεν μας άρεσε βέβαια. Αλλά παρόλα αυτά η απόφαση ελήφθη και η απόφαση την οποία θα πάρει το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ακολουθεί αυτή την πορεία. Τέλος, θα μπορούσαμε βέβαια να αλλάξουμε το μέγεθος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ότι καταλήξαμε σε 751 έδρες, δηλαδή 750 συν τον πρόεδρο όπως λέει η συνθήκη, είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη στα τελευταία 20 λεπτά της διακυβερνητικής. Ήμουν παρόν εκεί και ξέρω ποιος είναι ο υπεύθυνο και ξέρω ε, και τους λόγους για τους οποίους έγινε κάτι τέτοιο. Ήταν εντελώς αφαίρετο. Δεν υπάρχει καμία μαθηματική λογική πίσω από τον αριθμό 750 ή 751. Ή επίσης ε, και ε, δεν υπάρχει και καμία λογική τεκμηρίωση του αριθμού 96 για τη Γερμανία. Πέρα από την ιστορία γύρω από όλα αυτά βέβαια, τα οποία παραπέμπουν στο Μάστριχτ. Πολλά μένει να συζητηθούν λοιπόν. Περιμένουμε την τελική έκθεση από τον καθηγητή Γκρέμιτ και θα ήθελα για μια ακόμη φορά να τον ευχαριστήσω για την τεράστια προσπάθειά του και στο Κέμπριτζ και για την παρουσία του εδώ το απόγευμα στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Κύριο Χέφνερ έχει το λόγο πάλι. Ήθελα απλά να υπενθυμίσω. Ρωτήσατε κύριε καθηγητά το εάν απαντήσατε τις ερωτήσεις. Ε, δεν απαντήσατε στη δική μου. Δεν ξέρω γιατί. Θέλω να την ξαναθέσω. Ίσως μπορείτε να μου απαντήσετε γραπτός. Θέλω να, να ληφθεί υπόψη αυτή η ανησυχία. Σας ρώτησα ποιος θα ήταν ο διαιρέτης με το 6 και το 96 ως ανώτατο και κατώτατο όριο ως δεδομένα με έναν ενιαίο διαιρέτη να καταλήξουμε σε μια κατανομή με ευθύνουσα αναλογικότητα και να υπάρχει μια στρογγυλοποίηση. Και η απάντηση το ότι έπρεπε να χτίσουμε νέο κτίριο είναι λάθος μαθηματική. Είναι θέμα υπολογισμών. Το θέμα είναι ποιο θα ήταν αυτός ο διαιρέτης. Και ε, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας και θα την αναμείνω με, με αγωνία. Κύριε καθηγητά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να διατυπώσω την ερώτηση που έκανε που υπέβαλα και προηγουμένως. Δεν είναι ερώτηση μαθηματικού, είναι μια κοινότυπη ερώτηση. Λοιπόν, Λέγω, σύμφωνα με τις ηθίκες, ορισμένα κράτη πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα μήνυμο με έξι βουλευτών. Άσχετα αν μέσα από τους μαθηματικούς υπολογισμούς δεν καταφέρνουν να έχουν αυτό τον αριθμό των βουλευτών. Γιατί δεν δίνουμε κατευθείαν σε όλα τα κράτη-μέλη έξι βουλευτές και μετά Προχωράμε στον κλασικό υπολογισμό ε, σύμφωνα με την αναλογικότητα του πληθυσμού σε όλα, τα κράτη εκτός από εκείνους που πήραν αυτό το μίνιμουμ των 6. η Γερμανία σήμερα και αύριο κάποια άλλη χώρα θα μπορούσαν ίσως να, θα μπορούσαν τους αντιστοιχεί παραπάνω βουλευτές από αυτούς που έχουν σήμερα. Εμείς θα μπορούσαμε όμως να κάνουμε την αφαίρεση και πάει λέγοντας. Λοιπόν, να κρατήσουμε εμείς δηλαδή την αναλογία, να μην έχουν πάνω από 96 και να μην έχουν κάτω από 6. Και έτσι σεβόμαστε τους όρους. Για να πλουστεύσουμε λοιπόν τα πράγματα, μια χώρα με 10 εκατομμύρια κατοίκους θα πρέπει να έχει 6 φορές λιγότερους βουλευτές από τη χώρα εκείνη που έχει 60 εκατομμύρια. Είναι λάθος αυτός ο τρόπος σκέψης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ενθυμίστε ότι είχατε θέσει κι άλλο ένα ερώτημα το οποίο δυστυχώς δεν απάντησα. Το πώς το προτινόμενο σύστημα συμπεριφέρεται στην περίπτωση όπου ενταχθούν μεγάλες χώρες. Πολύ εύκολα είναι η απάντηση. Αν μια μεγάλη χώρα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν την Τουρκία σαν παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση αφαιρείται το ανώτατο των 96 γιατί η μεγάλη χώρα θα παίρνει πάρα πολλές έδρες οπότε όλα τα άλλα κράτη θα πρέπει να παραδώσουν έδρες και δεν βάζω την πρόπτικη αυτή γιατί έτσι κι αλλιώς όλες οι χώρες θα έχουν κάτω από 96 από μαθηματικής επόψεως λοιπόν η ένταξη μιας μεγάλης χώρας σαν την Τουρκία καθιστά την εφαρμογή της φόρμουλας αυτής απλούστερη και πιο λογική, ορθολογική καλύτερα. Για τον κύριο Χέφνερ, ζητώ συγγνώμη που δεν απάντησα στην ε, ερώτησή του. Προσπάθησα αλλά δεν το έκανα με σωστό τρόπο. Λέει γιατί δεν διαχωρίζουμε εμείς τις περιπτώσεις από το 6 μέχρι το 96. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Και θα έχετε σε αυτή την περίπτωση ένα μικρότερο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες και συγκεκριμένοι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και αν κάνει κανείς αυτό το διαχωρισμό, ακριβώς γιατί οι μεγάλες χώρες συμπιέζονται, όλες οι άλλες χώρες θα συμπιεστούν και αυτές. Αυτό είναι κάτι το οποίο δικαιολογείται σε επίπεδο αρχής, τεκμηριώνεται σε επίπεδο αρχής και σε επίπεδο αναλογικότητας είναι κάτι το οποίο φαίνεται πιο υπερασπίσιμο και ικανοποιητικό. Σε πάρα πολλές χώρες θα υπάρξουν απώλειες εδρών και το σύνολο του μεγέθους δεν θα είναι 751, θα είναι πολύ λιγότερο. οπότε δεν θα χρειαστείτε μεγαλύτερο κτίριο. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο αριθμός αυτός, μπορούμε να το υπολογίσουμε, δεν το έχουμε κάνει αυτό. Και δεν το έχουμε κάνει γιατί μας είπατε ότι θα πρέπει όσον αυτό είναι δυνατό να φτάσουμε τον αριθμό 751. Δεν ήταν καθοριστικός περιορισμός αυτός, ήταν επιθυμητός περιορισμός. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ποιος είναι ο διαιρέτης στη συγκεκριμένη περίπτωση, εσείς θα πρέπει να τον επιλέξετε, αλλά σίγουρα θα οδηγήσει ένας διαφορετικός διαιρέτης, ένα μικρότερο σώμα και κατά συνέπεια πάρα πολλές μεγάλες χώρες θα χάσουν έδρες. Κύριε Πρόεδρε, διορθώστε με αν κατάλαβα καλά. Ας προσπαθήσω να παραφράσω την ερώτησή σας. Να το κάνω αυτό, τον τρόπο με τον οποίο εκλέγεται, κατανέμονται οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Στη ΣΥΠΑ, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο αριθμός των εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι, και εδώ υπάρχει μια διατύπωση υποσυζήτηση, είναι αναλογικός με τον αριθμό των πολιτών κάθε πολιτείας. Ελάχιστος αριθμός είναι το ένα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα θέμα στρογγυλοποίησης το οποίο συζητιέται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι αντικείμενο πολλών πανεπιστημιακών μελετών. Πάντα χρησιμοποιείται ένας διαιρέτης, είναι απαραίτητο να υπάρξει ένας διαιρέτης για να ικανοποιηθούν οι περιορισμοί και υπάρχει αναλογική κατανομή με βάση αυτό τον διαιρέτη έτσι ώστε κάθε χώρα που έχει λιγότερο από ένα στον τελικό υπολογισμό να παίρνει ένα τουλάχιστον αντιπρόσωπο. Στην περίπτωση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ίδιο κάνουμε. Όποιος έχει λιγότερες από έξι θα φτάσει στις έξι. Αυτή είναι θα έλεγα μια βασική αρχή κατανομής των εδρών και είναι μία αρχή η οποία δεν εξυπηρετεί τελικά πάρα πολύ τις μικρές χώρες. Δεν θέλω να κάνω τώρα τις διαιρέσεις ε, ε, οι οποίες είναι ε, σχετικά περίπλοκες αλλά οι πράξεις δείχνουν ότι κάθε χώρα που δεν φτάνει επί πληθυσμιακής βάσεως 6 παίρνει 6. Οπότε σε αυτή την περίπτωση για να πάρεις 6 μπορείς να κάνεις τον απαραίτητο υπολογισμό. Δηλαδή αυτοί που αξίζουν τους 6 παίρνουν 6, αυτοί που δεν αξίζουν τους 6 πάλι παίρνουν 6. Οπότε οι μικρότερες χώρες εδώ θα έλεγα χάνουν σε σχέση με τον υπάρχοντα τρόπο κατανομής. Εμείς ερμηνεύσαμε τον δρόμο αυτό σαν έναν δρόμο που δεν σέβεται τη φήνουσα αναλογικότητα και γι' αυτό δεν περιλαμβάνεται στην πρότασή μας. Κοιτάξτε, ίσως δεν έχω απαντήσει πλήρως σε αυτά τα οποία ρωτήσατε. Ε, είμαι στην διάθεσή σας όποτε θέλετε. Για μένα είναι πολύ ευχάριστη η διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη των μελών της Επιτροπής. Είναι σαφές ότι αν κάποιος μας δώσει εξηγήσεις ή ζητήσει εξηγήσεις, από πού τα μάθαμε όλα αυτά θα του πούμε από το Cambridge. Νομίζω ότι θα κλείσουμε τη συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Θυμίζω ότι για να υπάρξουν τροπολογίες η προθεσμία Μαρτίου. των τροπολογιών είναι η 17η Μαρτίου. Εντάξει. Α, όχι, όχι, όχι Μαρτίου, Φεβρουαρίου, Φεβρουαρίου η προθεσμία. Θα πρέπει επίσης να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα που μας περιμένει. Ναι, λοιπόν, εμεί περιληπτικά έχουμε μια έκτακτη συνάντηση στι 14 Φεβρουαρίου από τι 8 μέχρι τις 9.30 στο Στρασβούργο. Ε. Α, άλλαξε. Ε, τότε πείτε, με, πείτε μου τι πρέπει να διορθώσω. Λοιπόν, υπάρχει ένα λάθος το οποίο τεκμηριώνει ένα άλλο λάθος. Στην πραγματικότητα η έκτακτη συνεδρίαση της 14 η θα είναι από τις 9 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. τέτοιου είδους ωράρια δημιουργούν ε, θα έλεγα σύγχυση. Μια επόμενη έκτακτη συνάντηση 17 Φεβρουαρίου από τις 10 ε, μέχρι τις 12. Επίσης έχουμε την επόμενη τακτική 14 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και την τρίτη που ακολουθεί 15 Μαρτίου από τις 9 μέχρι τις 12.30 στις Βρυξέλλες. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ε, λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση ούτε για τα ωράρια. Τώρα τελειώνουμε. Ευχαριστώ. Appunto, quindi è meglio